Καλησπέρα συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι. Έχουμε μαζί μας σήμερα την Εστονική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τρεις υπουργούς την κυρία Κάντρι Σίμψον, Υπουργό Οικονομικών και Υποδομών, υπεύθυνη και για θέματα ενέργειας και βιομηχανίας. Να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της Εστονικής Προεδρίας η Επιτροπή Ήτρε θα επεξεργαστεί πολλούς σημαντικούς φακέλους σε αυτούς τους τομείς πολιτικής, όπως είναι το πακέτο μέτρων για την καθαρή ενέργεια, κλητορικές επικοινωνίες, πρωτοβουλίες ε, σε, στον τομέα του διαστήματος και της άμυνας και θα ξεκινήσουμε και τις εργασίες μας για το πρόγραμμα για το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο. Η προετοιμασία δηλαδή. Όλα αυτά σχετίζονται με τα ζητήματα της βιομηχανίας, της ανταγωνιστικότητας και της ενέργειας. Επιτρέψτε μου να πω ότι διανύουμε μία περίοδο κατά την οποία θέλουμε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε κάποιες ε, ε, διαπραγματεύσεις σε ορισμένους ε, φακέλους τουλάχιστον και περιμένουμε από την Εστονική Προεδρία να καταλήξει σε κοινή θέση τουλάχιστον για, το, τη δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μας. Βεβαίως αυτό που ενδιαφέρει πολύ την Εστονική Προεδρία είναι το ψηφιακό θυματολόγιο καθώς η Εστονία είναι μία από τις καλύτερα προετοιμασμένες χώρες από αυτή τη σκοπιά. Περιμένουμε λοιπόν να ε, δεχθούμε την ειδική, μια ειδική, ιδιαίτερη μεταχείριση της Επιτροπής Ήτρε από την Αστωνική Προεδρία. Ε, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Παρακαλώ, έχετε την ευκαιρία να μας παρουσιάσετε τώρα το πρόγραμμα ε, της Αστωνικής Προεδρίας στις δικές σας αρμοδιότητες. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, επιφυλάσσουμε ειδική μεταχείριση στην Επιτροπή σας. Να πω και κάτι προσωπικά. Ε, ε Χαίρομαι πολύ που ξεκινούμε σε αυτό το ακαδημαϊκό ε, επίπεδο της συζήτησή μας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά και αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ε, Βιομηχανίας και Έρευνας, είναι μεγάλη μου χαρά ε, που βρίσκομαι εδώ μαζί σας για να συζητήσουμε μαζί σας τις προτεραιότητες μας ε, για το δεύτερο μισό του χρόνου. Τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε ε, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο όσον αφορά τη θέσπιση στόχων για την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχοντα αυτά κατά νου, χαίρομαι πολύ που έχουμε αυτέ τι ευκαιρίε για την ανταλλαγή απόψεων ω συνάδελφοι. Είχαμε ένα πολύ καλό ε, διάλογο ήδη πέρσι στο Ταλίν και εγώ επίσης είχα πολύ χρήσιμες συζητήσεις μαζί σας εδώ και στις Βρυξέλλες αλλά και αλλού. Μαζί πρέπει να επιδιώξουμε την εξέβρεση των καλύτερων λύσεων ε, προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη έχει κοινό έδαφος πάνω στο οποίο μπορεί να βασιστεί προκειμένου να αντιμετωπίσει επιτυχώς όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε καθώς και για να αξιοποιήσει τις πολλές δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας. Να συνεχίσω με την ενεργειακή πολιτική, έναν ε, ζωτική σημασίας κλάδο για την κοινωνία, όπου βρισκόμαστε στο μέσο μιας θεμελιώδους ε, αλλαγής μεταβαίνοντας προς μια πλήρως λειτουργική ενεργειακή ένωση. Βασικός στόχος της Εστονικής Προεδρίας στο δεύτερο εξάμεινο του 2017 ε, βεβαίως ε, επικεντρώνεται στην νομοθετική δραστηριότητα. Το Συμβούλιο θέλει να εξασφαλίσει ενεργειακή τροφοδοσία βάσει της αγοράς, να μειώσει την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ενέργειας και να ε, θεσπίσει μια μελλοντοστραφή κλιματική πολιτική δουλεύοντας πάνω στις τέσσερις, ε, στους τέσσερις τομείς ε, της ενεργειακής πολιτικής. Ε, διαμόρφωση και σχεδιασμός ε, της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, διακυβέρνηση ενεργειακής ένωσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα. Η Εστονία λοιπόν θα εξασφαλίσει την ποιότητα και την ισορροπία της ε, νομοθεσίας. Και βασιζόμενοι στο έργο της Μαλτέζικης Προεδρίας θα προδιώξουμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο, ιδίως στις προτάσεις του πακέτου για την καθαρή ενέργεια με ιδιαίτερη ε, ε, εστίαση στον επανασχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μια εύρυθμη λειτουργία της αγοράς είναι βασικός ε, κινητήρος μοχλός για την ανάπτυξη στην τροφοδοσία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καλός δείκτης για την ενεργειακή πολιτική. Η εξορθολογισμένη διακυβέρνηση για την πολιτική ενέργειας και κλίματος πρέπει να είναι το βασικό εργαλείο για την επίτευξη διατομιακών στόχων μακροπρόθεσμα και να μειώσει το διοικητικό άχθος. Σημαντικό στοιχείο, στοιχείο κλειδί θα είναι να ε, ενισχυθεί η διαφάνεια και η σαφήνεια στις πολιτικές μας. Κάτι που ε, ε, αναμένουν από εμάς επενδυτές και διεθνείς εταιρεία αλλά και η κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε δύο γύρους τριμερούς διαλόγου για τις προτάσεις για την ενεργειακή αποδοτικότητα με το Κοινοβούλιο. Και αναλόγω τη διαθεσιμότητα του Κοινοβουλίου, εμεί θα θέλαμε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις το αργότερο τον Νοέμβριο και να καταλήξουμε σε συμφωνία τουλάχιστον ω προ την οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων ψηφιακή προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οριζόντια προτεραιότητα σε όλους τους ε, κλάδους και τομείς και συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς, σε αυτούς τους τομείς βεβαίως και ο κλάδος ενέργειας. Θα ε, συνεργαστούμε λοιπόν με τα κράτη-μέλη προκειμένου να εκδοθεί μια διακήρυξη σχετικά με τις ε, συνέργειες που μπορούν να υπάρξουν στον τομέα των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επίσης, όσον αφορά το Nord Stream 2, θα ξεκινήσουμε συζητήσεις σχετικά με τη σύσταση τη για τη διαπραγμάτευση τη εντολή στη διάρκεια τη Προεδρία μα. Η πρώτη συζήτηση προγραμματίζεται να γίνει στι 25 Ιουλίου. Περνώντα τώρα από την ενέργεια σε άλλα θέματα, πρέπει να σα πω ότι είμαι αρμόδια και για ζητήματα ανταγωνιστικότητα. Ε, μιλώ για την ε, βιομηχανική πολιτική. Στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας του Μαΐου όλα τα κράτη-μέλη προσαφήνισαν ότι ο κλάδος της βιομηχανίας και της μεταποίησης θα πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες ε, πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό επισημάνθηκε και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη σύνοδό του Ιουνίου. Το Συμβούλιο κάλεσε την Κομισιόν να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια βιομηχανική στρατηγική και να παρουσιάσει στρατηγικούς στόχους για τη βιομηχανία. Επίσης ζήτησε να καταρτιστεί ένα σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα μέτρα. Χαιρετίζουμε επίσης το ψήφισμα σχετικά με τη βιομηχανική στρατηγική που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα η Εστονική Προεδρία υποστηρίζει πλήρω όλα αυτά τα αιτήματα του Κοινοβουλίου και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Στη διάρκεια τη Προεδρία μα θα επικεντρωθούμε και στο ζήτημα τη ψηφιοποίηση, τη βιομηχανία και τη ε, προηγμένη μεταποίηση. Γνωρίζουμε ότι είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό για το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα για τη δική σας Επιτροπή. Καθώς μιλούμε για την βιομηχανία, θα ήθελα επίσης να εκφράσω την υποστήριξή μας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αμυντικής Βιομηχανίας και ελπίζουμε ε, στην, να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό το τελευταίο. Χαιρόμαστε λοιπόν που έχουμε το Κοινοβούλιο ως εταίρο σε αυτή τη διαδικασία, ιδίως έχοντας κατά νου το ψήφισμα του Νοεμβρίου του 2016, με το οποίο καλείται η Κομισιόν να ενισχύσει τη βιομηχανική και τεχνολογική βάση του αμυντικού τομέα. Καθώς η Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία είναι ζωτική σημασίας και απασχολεί μισό εκατομμύριο άτομα, ελπίζουμε οι φάκελοι αυτοί να προχωρήσουν γρήγορα. Να πω και δύο λόγια για την πρωτοβουλία για τις νεοφυείς και τις επεκτηνόμενες επιχειρήσεις. Το δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να, ε, στο οποίο θέλω να επικεντρωθούμε είναι ε, οι νοφεί και επεκτηνόμενες επιχειρήσει. Όπω γνωρίζετε, το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα χαιρέτησε τη σχετική πρωτοβουλία τη Κομισιόν και το Συμβούλιο υποστηρίζει πλήρω αυτή την προσέγγιση που προτάθηκε να ακολουθηθεί σχετικά με την ανάπτυξη ενό καλύτερου περιβάλλοντος για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα που θα βοηθά στη δημιουργία και την επέκταση των νεοφυών επιχειρήσεων. Η Εστονική Προεδρία ε, σκοπεύει να δώσει συνέχεια σε αυτήν την πρωτοβουλία της Κομισιόν και κατά τη διάρκεια της θητείας μας θα προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί καθώς και για ε, την, ε, τις δράσεις που είναι αναγκαίες για τα επόμενα χρόνια. Και με αυτά θα ήθελα να κλείσω την παρέμβασή μου. Είμαι βεβαίως ε, στη διάθεσή σας ε, ε, για ερωτήσεις σχετικά με ζητήματα που άπτονται της βιομηχανίας και της ε, καινοτομίας. Οι άλλοι συνάδελφοι που είναι μαζί μας θα καλύψουν τα υπόλοιπα θέματα. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων να πάρουν το λόγο και να σχολιάσουν. Η κυρία Δελκαστήγιο νομίζω, εκ μέρους του ΕΛΚ, ο λόγος είναι δικό σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Να σας πω πως ήταν ιδιαίτερα θετικό το ότι είχαμε τη δυνατότητα να σας ακούσουμε για τη δέσμευση που έχετε αναλάβει στον κλάδο της ενέργειας και νομίζω ότι είναι ένα από τα πολύ μεγάλα ζητήματα τα οποία αφορούν πια την Επιτροπή μας. Ξέρετε πως έχουμε και άλλα ε, θέματα τα οποία μας απασχολούν, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε το πακέτο για την καθαρή ενέργεια και νομίζω ότι αυτό είναι ίσως και το πιο κομβικό ε, θέμα από αυτά που συζητάμε. Πιστεύουμε πως ε, κατά τους επόμενους μήνες μετά το καλοκαίρι θα καταφέρουμε τουλάχιστον να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση στο Συμβούλιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεράσουμε αυτό το σημείο, αλλά τουλάχιστον αυτό θα το επιδιώξουμε. Και να σας πω ότι η δική μου προσωπική άποψη, και θα επιμείνω σε αυτό, είναι πως υπάρχουν δύο βασικά σημεία τα οποία σχετίζονται περισσότερο με την διακυβέρνηση όπως επίσης και ο σχεδιασμός της νέας εσωτερικής αγοράς για την ηλεκτρική ενέργεια. Θέματα τα οποία σχετίζονται και με τις δυνατότητες διασύνδεσης και τους κόμβους ε, βρόχους διασύνδεσης. Να σας πω πως η χώρα μου επηρεάζεται, όπως και άλλες, και θα θέλαμε να προχωρήσουμε έτσι ώστε να αποκτήσουμε μια νέα αγορά για την ενέργεια και για να καταφέρουμε κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο όλα τα κράτη-μέλη να βρουν τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η διασύνδεση που είναι απαραίτητη. Άρα λοιπόν οι συγκεκριμένοι στόχοι θα πρέπει να ενισχυθούν όχι με υψηλότερα ποσοστά της ηλεκτρικής ενέργειας που υπάρχει σε κάθε χώρα, τα οποία θα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένα, αλλά βρίσκοντας τον τρόπο με τον οποίο αν αναλύσουμε τη σχέση κόστους-οφέλους, θα γίνει συμφέρουσα η επένδυση σε αυτούς τους βρόχους διασύνδεσης. Και νομίζω ότι εξαρτάται μετά από κάθε κράτος μέλος τι θα κάνει τώρα. Να σας πω πως αυτή είναι και η άποψη της ομάδας του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Από τους σοσιαλιστές, ο κύριος Ζωρίνιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την ε, κυρία Υπουργό και να της ευχηθώ κάθε επιτυχία στην ε, Προεδρία της Εστονίας από την οποία έχουμε πολλές προσδοκίες και να σας πω πως ε, κυρίως στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ε, ψηφιακή ένωση. Και δεδομένου του γεγονότος πως στη χώρα της, στο χώρο αυτό, οι επιδόσεις τους είναι άριστες, να δούμε πώς μπορούμε και εμείς να χρησιμοποιήσουμε όσο δεν τον περισσότερο αυτές τις νέες τεχνολογίες. Έχουμε εδώ και μετά τους υπουργού Παιδείας, Επιχειρηματικότητας και νομίζω ότι το γεγονός που συγκεντρωθήκατε έτσι είναι πολύ συμβολικό. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ενιαία ψηφιακή αγορά που δημιουργεί μια ψηφιακή ένωση. Για να είμαστε πετυχημένοι θα πρέπει να έχουμε τεχνολογία εχμής, θα πρέπει να δημιουργήσουμε πλούτο και θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη ε, το πώς μπορούμε να ανοίξουμε τις πόρτες σε όλους τους πολίτες, έτσι όλοι να μπορέσουμε να δρέψουμε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η κοινωνία της πληροφορίας. Εσείς με πολλές λεπτομέρειες μας πήγατε ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες και θα εστιάσω σε δύο σημεία. Καταρχήν, να σας πω πως είμαι εισηγητής ε, στην πρωτοβουλία του Wi-Fi for You, δηλαδή η τοπική διασυνδεσιμότητα, το οποίο είναι κάτι ελπίζουμε θα κλείσει υπό τη δική σας προεδρία και είναι κάτι το οποίο έχει ένα τεράστιο δυναμικό. Δηλαδή, να έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ από δημόσιους χώρους. Και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει την εξάπλωση κοινωνίας πληροφορίας στην Ευρώπη. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν εσείς η Εστονική Προεδρία αυτή τη δυνατότητα θα τη χρησιμοποιήσετε γιατί είναι κάτι το οποίο ως πρωτοβουλία θα αρχίσει να τρέχει αυτό το εξάμεινο. Επίσης κάτι το οποίο φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι η πρόθεση να υπάρχει αυτή η διασταύρωση μεταξύ ψηφιακού και ενεργειακού στα πλαίσια του πακέτου για την ενέργεια. Γιατί νομίζω πως η υπηρεσία της πληροφορίας θα πρέπει να μπει στην, και να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των όσων συμφωνήθηκαν στο Παρίσι. Δηλαδή ο συνδυασμός ψηφιακών δικτύων με ενεργειακών δικτύων και αυτό θα μας δώσει ένα επιπλέον πλεονέκτημα που θα μας κάνει πιο ανταγωνιστικούς στην βιομηχανία, στις υπηρεσίες, παντού. Όλοι λοιπόν έχουν πάρα πολλές προσδοκίες από τη δική σας Προεδρία και πιο συγκεκριμένα στα δύο αυτά θέματα. Να δούμε δηλαδή, απαντήστε μου, τι θα γίνει με το Wi-Fi for You, θα το χρησιμοποιήσετε και πώς θα κάνετε αυτό το συγκερασμό ενέργειας και ψηφιακού. Ο κύριος Δανάουσκη έχει το λόγο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας κυρία Υπουργέ και νομίζω πως η δική σας Προεδρία φτάνει μια στιγμή όπου συζητάμε ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που μας αφορούν. Και αυτό είναι το ενεργειακό πακέτο, το οποίο θα επηρεάσει τις οικονομίες μας για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Ξέρετε πως η οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλα τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ενεργειακά θέματα. Μας είπατε πως θα γίνουν δύο τριμερείς διάλογοι, οι οποίοι θα καλύψουν τα θέματα αυτά. Και εκεί έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση να σας κάνω. πώς θέλετε να διατηρηθεί η συνέπεια και η συνοχή μεταξύ αυτών των επτά θεμάτων και χώρων που μας απασχολούν. Για παράδειγμα, ενεργειακή αποδοτικότητα. Πώς θα το προωθήσετε μέσω του Συμβουλίου. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές απόψεις, πολλές διαφορετικές προσδοκίες, πολλές αντικρουόμενες ματιές. Οπότε ξέρω πως ζητώ την προσωπική σας άποψη, αλλά πείτε μου ποιες είναι οι προσδοκίες σας, για παράδειγμα, για την αποδοτικότητα. Ευχαριστώ. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να μιλήσω εστονικά, οπότε θα τα πω στα εστονικά. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες τις ερωτήσεις και να μιλήσουμε για τον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Συζητήσαμε τα θέματα αυτά στην Επιτροπή μας και μιλήσαμε πάρα πολύ για θέματα σχεδιασμού και είναι κάτι το οποίο για μένα είναι σαφές. Και φαίνεται πως πολλοί από εμά δεν πιστεύουν πως αυτό που πρέπει να προκρίνουμε είναι μια προσέγγιση που θα βασίζεται στις αγορές. Άρα λοιπόν, το αντίστοιχο θέμα, πώς το συζητάτε στο Συμβούλιο, τι πιστεύετε. Ελπίζετε πως θα κλείσει μια συμφωνία για το πώς θα σχεδιάσουμε την ενεργειακή μας αγορά, την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, πώς θα λειτουργεί καλύτερη ιστορία αγορά ενέργειας. Να σας πω πως και για μας είναι μια ε, πρώτη εμπειρία να σας ακούμε να μιλάτε εστονικά. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Τούρμες. Θα μιλήσετε κι εσείς εστονικά. Αν μιλήσω εστονικά δεν θα πω πολλά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ και σας ευχαριστώ που μάλιστα μας υποδέχεστε στις 29 Σεπτεμβρίου στην Προεδρία που έχετε για τη Βαλτική πλέον γίνεται η πρώτη 100% ΑΠΕ περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να σας και κάθε επιτυχία για όλα τα υπόλοιπα. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο περισσότερα για την περιφερειακή συνεργασία με πρακτικά λόγια, είστε μία από τις περιφέρειες οι οποίες ε, είχατε τα μεγαλύτερα αποτελέσματα από τη ζεύξη με άλλες αγορές. Οπότε, ποια είναι η εμπειρία σας. Και δεύτερον, με κάπως πως στο μνημόνιο κατανόησης για την απεξάρτηση, από συγχρονισμό από το ρωσικό σύστημα και τον συγχρονισμό με το ευρωπαϊκό δεν έχει υπογραφεί ακόμα. Οπότε ήθελα να σας ρωτήσω γιατί. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να έχουμε τρεις βαλτικές χώρες οι οποίες τραγουδούν στον ίδιο ρυθμό. Είστε έτοιμοι? Είστε έτοιμοι να κάνετε παιχνίδι μαζί? Και επίσης για τη βιομηχανική πολιτική, κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας, νομίζω ότι θα ε, φτάσει και μια καινούρια ε, πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αυτοκίνητα, γιατί και η αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει να κάνει κινήσεις, γιατί διαφορετικά οι Κινέζοι θα κατακτήσουν και αυτό το κομμάτι της βιομηχανίας μας. Έχετε λοιπόν στρατηγική για το τι κίνητρα θα δώσετε στην αυτοκινητοβιομηχανία και τις κυβερνήσεις για να προλάβουν αυτές τις ε, τεχνολογικές επαναστάσεις που περιμένουν στον κλάδο τους. Uh, uh of... Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ήθελα εγώ να καλησορίσω εδώ την Υπουργό. Ε, και βέβαιως να της ε, ευχηθώ δύναμη. Γνωρίζω εκ πείρας πόσο δύσκολο είναι ε, μια μικρή χώρα να προεδρεύει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ κατάγομαι από την Κύπρο ε, και πριν από πέντε χρόνια είχα αυτή την ιδιότητα να προεδρώσω κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας και ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Εύχομαι κάθε επιτυχία και δύναμη πάνω απ' όλα. Το άλλο που ήθελα να ρωτήσω, ανεβερθήκατε για στον επανασχεδιασμό της αγοράς. Όμως, τα τελευταία χρόνια γίνεται μια συζήτηση γύρω από τα θέματα της απομόνωσης κρατών και περιοχών από τα μεγάλα ενεργειακά δίκτυα, διότι υπάρχουν ακόμα και κρατημένοι και περιοχές που είναι απομονωμένα από τα ενεργειακά δίκτυα. Το τι θα γίνει μέσα σε αυτόν τον σχεδιασμό στη βάση της Ενεργειακής Ένωσης. Το δεύτερο είναι η ενεργειακή φτώχεια. Είναι ένα νέο φαινόμενο που αγγίζει την Ευρώπη. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια εμείς στο Κοινοβούλιο να το τονίζουμε από την Επιτροπή να υπάρχουν μόνο διακηρύξεις, κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο ή συγκεκριμένα μέτρα για αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου που ένα και περισσότερο επηρεάζει εκατομμύρια πολίτες στην Ένωση. Το τρίτο αναφερθήκατε στη μείωση της ε, εξάρτησης και στο Nord Stream 2. Όμως δεν άκουσα κάτι να γίνεται σε σχέση με, την νότια, με τον νότιο αγωγό, την νότια Ευρώπη, που έχει μεγάλα προβλήματα στην ενεργειακή τροφοδεσία. Και ακόμα ένα ερώτημα, ξέρω τις επιτυχίες που έχει η Εσθονία, τα είπε και ο συνάδελφος ο Κλώτ, σε ό,τι αφορά τη ΣΑΠΕ. Ε, Όμω ε, θα ήθελα, είπε, είπετε ότι στηρίζεται τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, αλλά θα ήθελα μια τοποθέτηση σε ό,τι αφορά του στόχου για τη ΣΑΠΕ και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Διότι η Επιτροπή τελικά μείωσε ακριβώ του στόχου που έχει θέσει το Κοινοβούλιο και ο τελευταίο, επειδή χαιρετήσετε τη στροφή ή την απόφαση που γίνεται για την αμυντική βιομηχανία, ε, θα ήθελα ένα σχόλιο πώ αντιμετωπίζω το φαινόμενο ότι μια μεγάλη περιοχή τη Ένωση, ιδιαίτερα η Νότια Ευρώπη, αντιμετωπίζει μια διαδικασία αποβιομηχανοποίηση ε, ω αποτέλεσμα τη κρίση και τη ύφεση. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ευχαριστώ και τώρα παρεμβάσει ενό λεπτού, κύριε Πέτεσεν. Ευχαριστώ. Να καλωσορίσω και εγώ την Υπουργό. Όπως είπαν και οι άλλοι συναδελφοί, περιμένουμε πολλά. Δύο ώρα για μόνο για τα θέματα της ενέργεια. Δεδομένων των φιλοδοξιών της επερχόμενης Προεδρίας, της Νέας Προεδρίας, ε, δεν ξέρω, μου φαίνονται πολύ φιλόδοξο όλα αυτά. Ελπίζω να τα πετύχετε. Και δεν ξέρω αν μπορείτε να περάσετε όλα αυτά από το Συμβούλιο στο τέλο τη χρονιά. Οπότε πείτε μα λίγο παραπάνω, πώ θα τα πετύχετε όλα αυτά πραγματικά. Είναι καλό να έχει κανείς φιλοδοξίε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να σα βοηθήσει. Αλλά να είμαστε και ρεαλιστέ. Θα θέλαμε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση από εσά. Συνεχίστε να είστε φιλόδοξοι, παρακαλώ, αλλά πείτε μα και ρεαλιστικά τι πρέπει να περιμένουμε. ευχαριστώ. Μπένσεν. Πρόεδρε, καλώς ορίζω και εγώ τις Υπουργούς και εγώ για την ενεργειακή πολιτική. Γνωρίζουμε ότι μια απελευθερωμένη ενεργειακή αγορά είναι καλή για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Όμως, όταν ακούω τις προσεγγίσεις των Υπουργών στο Συμβούλιο, Βλέπω ότι συμφωνούν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων για την ε, Ενεργειακή Ένωση. Διαβάζω τα συμπεράσματα των τελευταίων συμβουλίων, ε, αλλά φοβάμαι ότι δεν υπάρχουν αρκετές φιλοδοξίες. Γνωρίζουμε την εξάρτησή μας σε αέριο από τον κύριο Πούτιν και την εξάρτησή μας ε, σε ορεικτά καύσιμα από τη Μέση Ανατολή. Και υποτίθεται ότι προσπαθούμε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας για το καλό των μικρομεσαίων και ούτω καθεξής. Και την ίδια στιγμή γινόμαστε μάρτυρες ε, εθνοκεντρικών προσεγγίσεων από τους υπουργού. Βλέπουμε και πώς κινούνται οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς. Πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερη περιφερειακή συνεργασία. Χρειάζεται να επανεσχεδιαστεί η αγορά, όντως. Αλλά εκεί οι φιλοδοξίε φοβούμε ότι είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τι θα κάνετε λοιπόν Πώ θα εξασφαλίσετε μια πιο θετική, πιο δυναμική προσέγγιση από το Συμβουλίο Μπουρικόφερ. Πρόεδρε, δύο ερωτήσει όσον αφορά τη βιομηχανική πολιτική. Πρώτον, στην τελευταία λομέλεια, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με συντριπτική πλειοψηφία, ζητώντας μια ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική, την οποία θα προάγει βεβαίω το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Τι θα γίνει για την υλοποίηση αυτού του θεματολογίου. Δεν άκουσα τίποτα σχετικό, ούτε διάβασα κάτι στο πρόγραμμά σα. Δεύτερον, όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία, από το 2009 υπάρχει η οδηγία περί αμυντικών προμηθειών, η οποία δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Αν εφαρμοζόταν, θα γλιτώναμε δισεκατομμύρια σε κονδύλια τα οποία δαπανούν τα κράτη-μέλη γιατί δεν συμμορφώνονται με τους ελάχιστους κανόνες ανταγωνισμού στην αγορά. Τι θα κάνετε ώστε να εφαρμοστεί επιτέλους αυτή η οδηγία από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Το ερώτημά μου πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση με εκείνο του κυρίου Μπουτικόβα. Σε πάρα πολλά ψηφίσματα εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε τοποθετηθεί σε σχέση με την ανάγκη κατάρτισης μιας ολοκληρωμένης βιομηχανικής στρατηγικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ο κύριος Μποτικόβα ε, είχε συντάξει μια έκθεση και ένα ψήφισμα μάλλον για τις, για τις επικοινωνίες, εγώ για τους ιδιοδρόμους και πρόσφατα ε, ο κύριος Μπούζεκ έλαβε και μια επιστολή από 15 προέδρους ομοσπονδιών ε, κλαδικών και θέλω να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό μπορείτε εσείς να μας υποστηρίξετε σε αυτή τη διαδικασία ώστε να ασκήσουμε πίεση στην Κομισιόν επιτέλους να ε, προτείνει μια ολοκληρωμένη πολιτική στον τομέα της βιομηχανίας τουλάχιστον με τη μορφή μιας κάποιας ανακοίνωσης. Ευχαριστώ. Και μια σύντομη ερώτηση από μένα, λέει ο Πρόεδρος. Σύμφωνα με αναφορές ε, του τύπου, ε, η Εσωμική Προεδρία θέλει να διευρύνει την εντολή για, ε, για να, να καταρτήσει ένα νέο νομικό πλαίσιο για τον Nord Stream 2. Θέλετε να διευρύνετε την εντολή και σε άλλους εταίρους υπεράκτιους. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες προφορίες σχετικά με τις προθέσεις σας σε αυτό το τομέα, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας, καθώς είμαστε υπεύθυνοι βεβαίως για την εντολή αυτή και μελλοντικά φυσικά και για την συμφωνία ε, που ενδεχομένως ε, θα συναυθεί. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Ήτρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το μεγάλο φάσμα ερωτήσεων που μου θέσατε Γνωρίζω πολύ καλά ότι κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις θα ήταν καλύτερο να απαντηθούν από τις συναδέλφους μου. Εγώ βεβαίως θα κάνω ό,τι μπορώ. Βλέπω ότι υπάρχουν πολλά ερωτηματικά σχετικά με το αν θα είμαστε αρκετά φιλόδοξοι ή αρκετά ρεαλιστές. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε και τα δύο. Φιλόδοξοι και ρεαλιστές. Αλλά να ε, αδράξω και εγώ την ευκαιρία να μιλήσω εστονικά και να πάρω παράδειγμα από την ε, συνάδελφο Κάλλας, ε, μιας και έχουμε διερμηνείς στη διάθεσή μας. Άκουσα λοιπόν το ερώτημά σας και με ρωτήσατε για το τι θα επιτύχει η Εσθονία στον τομέα του πακέτου για την καθαρή ενέργεια. Είναι πολύ μεγάλο το πακέτο αυτό. Προβλέπονται δύο τριμερείς ε, διάλογοι για, την, ε, ε, για τα δύο αυτά σημαντικά έγγραφα. Μάλιστα καταλήξαμε σε κοινή θέση και στις 26 Ιουνίου, οπότε εμείς ως Συμβούλιο είμαστε, είμαστε έτοιμοι, έχουμε καταλήξει σε θέση. Θεωρούμε την ενεργειακή αποδοτικότητα είναι πραγματικά ε, πολύ σημαντικό θέμα. Η Εστονία λοιπόν έχει προχωρήσει ε, και έχει ε, συγκεκριμένο σχέδιο για όλα τα πακέ, όλα τα μέτρα, για όλες τις προτάσεις του πακέτου για την καθαρή ενέργεια. Έχουμε ήδη προγραμματίσει συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας και αυτό αφορά και την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης είναι ο βασικός στόχος που έχουμε θέσει και συνδέεται και με όλες τις νομοθετικές προτάσεις σχετικά που, που εντάσσονται στο πακέτο για την καθαρή ενέργεια. Αυτό το, αυτό το σύστημα διακυβέρνησης θα πρέπει να αποτελέσει το πλαίσιο το οποίο θα είναι και ισχυρό και ευέλικτο και που θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τους στόχους που έχουμε θέσει έως το 2030. Θέλουμε να μειώσουμε το διοικητικό άχθος και να παρακολουθούμε επίσης την πρόοδο που ε, σημειώνεται με το μικρότερο δυνατό διοικητικό ε, άχθος. Η κυρία Κάλλας λοιπόν έθεσε ένα ερώτημα σχετικά με το σχεδιασμό της αγοράς ε, ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ, στο οποίο έχουμε επενδύσει πολύ, στο οποίο έχουμε καταβάλει πολύ μεγάλες προσπάθειες, σχετικά με να, ε, προκειμένου να καταστήσουμε εύρυθμη τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά αποτελέσματα δεν μπορεί κανείς να περιμένει ενιανικτή. Η Εστονία θεωρεί ότι τέσσερις προτάσεις είναι πολύ σημαντικές σχετικά με το σχεδιασμό της Ενεργειακής ε, ε, Ένωσης. Θέλουμε να καταλήξουμε σε θέση του Συμβουλίου το Σεπτέμβριο. Ελπίζουμε ωστόσο το Κοινοβούλιο να παράσχει σε εμά την υποστήριξή του προκειμένου να καταλήξουμε σε τελική συμφωνία εντός του 2018. Υπήρξε επίσης ένα ερώτημα σχετικά με την πρωτοβουλία της Εστονίας ε, στον ψηφιακό κόσμο. Η συνάδελφος Ουρβεπάλο θα μιλήσει για αυτά τα θέματα και θα επικεντρωθεί μάλιστα σε αυτά. Όσον αφορά ωστόσο την, ε, τον ψηφιακό κόσμο και τον τομέα της ενέργειας, Πρέπει να σας πω ότι έχουμε σκοπό να καταλήξουμε σε διακήρυξη σχετικά με τις συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα και εκεί γίνεται αναφορά και στην ψηφιακή οικονομία και στα ζητήματα της ενέργειας. Μιλούμε για, την, ε, για το μέλλον του κλάδου της ενέργειας, για πλατφόρμες ανταλλαγής δεδομένων, για τους παραγωγούς και τους προμηθευτές με σκόπο να παρέχονται περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες στους καταναλωτές. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα απλό και υποστηρικτικό νομοθετικό πλαίσιο. Θέλουμε να έχουμε έξυπνους μετρητές οι οποίοι θα ε, λειτουργούν ε, από κοινού, θα είναι διαλειτουργικοί και ε, καμία συνεδρίαση υπό Προεδρία δεν θα αγνοήσει ε, αυτό το ζήτημα των ε, ψηφιακών πλατφορμών. Σας διαβεβαιώ. Κάποια μέλη της Επιτροπής έθεσαν ερωτήματα σχετικά με την Εστονία. Ο κύριος Τούρμες ρώτησε για την πρόοδο της Εστονίας όσον αφορά τον αποσυγχρονισμό της Εστονίας και των γειτόνων, των γειτονικών κρατών είναι αλήθεια ότι είμαστε συγχρονισμένοι στο ίδιο δίκτυο με Ρωσία και Λευκορωσία. Και θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Έχουμε μάλιστα εξετάσει και αναλύσει διάφορα σενάρια στο Συμβούλιο όσον αφορά τον αποσυγχρονισμό μας από το ρωσικό και λευκορωσικό δίκτυο. Υπάρχουν πολλές ανοιχτές ε, πιθανότητες, όμως δύο, ε, δύο είναι οι βασικές μας ε, γραμμές εστίασης αυτή τη στιγμή. Μία είναι ο, ο διάδρομος που θα οδηγεί μέσω Πολωνίας. Πάντως, έως το τέλος της χρονιάς Ελπίζουμε να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, να έχουμε καταλήξει σε ορισμένες ε, λεπτομέρειες, ε, να έχουμε στη διάθεσή μας και τις σχετικές μελέτες ώστε να οδηγήσουμε, να οδηγηθούμε και σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Ο πρόεδρος μίλησε για το Nord Stream 2. Πράγματι, θέλουμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις για την εντολή για τον αγωγό Nord Stream 2 το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, οι Υπουργοί Ενέργειας συνεδρίασαν ε, στις 26 Ιουνίου και το θέμα αυτό ε, συζητήθηκε μόνο ως ενημερωτικό σημείο. Δεν έχει υπάρξει ακόμα έγκριση κάποια συγκεκριμένης προσέγγισης. Η τυπική συζήτηση, η ουσιαστική συζήτηση μάλλον θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου επί του θέματος αυτού. Εμείς έχουμε πολλές φιλοδοξίες. Θέλουμε να ακούσουμε και από τα κράτη-μέλη ποια είναι η δική τους γνώμη, ποιες είναι οι δικές τους απαιτήσεις σχετικά με τον, με τον τρίτο αγωγό και ε, ε, πρέπει να καταλήξουμε για το αν η διαπραγμάτευση θα γίνει μόνο για τον Nord Stream 2 ή, και, ή αν θα συμπεριλαμβάνει και μελλοντικού αγωγού και τον South Stream. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα τι γνώμε των κρατών μελών και στη συνέχεια θα καταλήξουμε σε, σε θέση. Γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει ευρύτατη κατανόηση του νομικού πλαισίου που θα καταρτήσουμε το οποίο με τη σειρά του θα μας δώσει τη δυνατότητα να ερμηνεύσουμε τις, ε, τους διάφορους τρόπους αξιοποίησης αλλά και τις δυνατότητες που ε, ανοίγονται εν ώψη της κατασκευής αυτών των αγωγών και ποιες δυνατότητες ανοίγονται για την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να προχωρήσει στο στόχο της διαφοροποίησης για την βιομηχανική στρατηγική θα συνεχίσουμε τη συζήτηση επί του θέματος αυτού. Θέλουμε να καταρτήσουμε, να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο μέσω του οποίου θα ορίζονται οι διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα αφορούν την ψηφιοποίηση, τη βιωσιμότητα, τις νεοφυείς ε, επιχειρήσεις, και τα λοιπά. Θέλουμε λοιπόν να ε, υποβάλει η Κομισιόν μια πρόταση για στρατηγική έως τον Απρίλιο του 2018 όπως μάλιστα αναφέραμε ρητός και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να εργαστούν επί μιας τέτοιας στρατηγικής, σας διαβεβαιώ. Ευχαριστώ πολύ. Εκτός μικροφώνου. Δεν είναι πάντα εύκολο να συγκεντρώσει κανείς όλες τις ερωτήσεις. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε. Έχουμε μία οδηγία για τις κρατικές προμήθειες, η οποία ψηφίστηκε το 9 και η οποία περιγράφει τα πρότυπα που πρέπει να ακολουθούμε στις συμβάσεις για την άμυνα, τις αμυντικές κρατικές προμήθειες, που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Η ερώτησή μου είναι, η Προεδρία σας θα ασχοληθεί με την εφαρμογή έτσι ώστε να έχουμε μία εξοικονόμηση πολύτιμων ε, χρημάτων των φορολογουμένων, τα οποία αυτή τη στιγμή σπαταλώνται. Thank you for Well, we will... Ευχαριστώ πολύ που το επαναλάβατε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε. I hope that will be enough. Ελπίζω να φτάσει λοιπόν αυτό, λέει ο μιλητής. Είδατε λοιπόν πως οι ερωτήσεις που σας έχουν απευθυνθεί είναι εξαιρετικά λεπτομερείς και είμαι σίγουρος πως η Εστονική Προεδρία όλα αυτά τα ερωτήματα θα τα μεταφέρουν πίσω στο Τάλιν και θα προσπαθήσουν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες σας. Λυπάμαι, συνάδελφα, αλλά πρέπει να πω το εξή. Αλλά το να μπούμε σε τέτοιε λεπτομέρειε αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο και δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανεί μέσα σε λίγα λεπτά. Όμω οι απαντήσει σα ήταν εξαιρετικέ. Μια πολύ ωραία παρουσίαση στην αρχή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το πόσο δεσμευμένοι είσαστε και σα εύχομαι καλή επιτυχία του επόμενου έξι μήνε που είναι τόσο σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε τώρα να περάσουμε σε ένα ακόμα θέμα που είναι η ψηφιακή, ε, το ψηφιακό θεματολόγιο, η τεχνολογία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε μαζί μας την Υπουργό κύριο Πάλο, η οποία είναι υπεύθυνη για τα θέματα αυτά, για την επιχειρηματικότητα και για την τεχνολογία της πληροφορικής. Κυρία Υπουργέ, είμαστε εδώ και με χαρά Περιμένουμε να σας ακούσουμε, να μας πείτε κι εσείς ποιο είναι το πρόγραμμά σας για το επόμενο εξάμεινο. Ξέρω πως δεν σας έδωσα πολύ χρόνο για να προετοιμαστείτε. Έτσι όμως θα προχωρήσουμε κι εμείς. Και είναι πολύ σημαντικό και να σημειώσετε όλες τις ερωτήσεις και κάποιες λεπτομερεί απαντήσεις γραπτά να τις στείλετε ε, στους συναδέλφους και βεβαίως να τα θυμόσαστε όλα αυτά κατά τη διάρκεια της προηγίας. Κυρία μου, θα ήθελα να μας πείτε ποιο είναι το πρόγραμμά σας. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ καθηγήτρια κυρία Μπούζεκ, μέλη της Επιτροπής κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ ευχαριστημένη που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας τις προτεραιότητες της Εστονικής Προεδρίας του Συμβουλίου παρόλο που δεν έχουν περάσει ούτε δύο εβδομάδες που έχει ξεκινήσει, μπορώ να πω πως εμείς εκτελούμε τα καθήκοντά μας ως Προεδρία και επίσης πως έχουμε αναλάβει δράση με μεγάλη αποφασιστικότητα. Πιστεύουμε πως η Ευρώπη έχει πάρα πολύ μεγάλο κοινό παρανομαστή που θα επιτρέψει με επιτυχία να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις που υπάρχουν σήμερα και να χρησιμοποιήσουμε στο μέγιστο τις δυνατότητε που προσφέρονται. Είμαι υπουργό για την τεχνολογία τη πληροφορίας και οι προκλήσεις και οι δυνατότητες που έχουμε στο χώρο της ψηφιοποίησης και του ψηφιακού κόσμου μου είναι θέματα ιδιαίτερα προσφυλή και θα ήθελα σήμερα να εστιάσω στα θέματα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία στην Επιτροπή Ήτρε. Μία από τις βασικές προτεραιότητες της Προεδρίας μας είναι να προωθήσουμε την ψηφιακή Ευρώπη μαζί με τους ε, εταίρους μας από το τρίο Προεδριών. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι το Συμβούλιο να σεβαστεί την προθεσμία για να κλείσει τις σχετικές διαπραγματεύσεις για όλους αυτούς τους ε, ε, φακέλους το 2018. Επίσης βασιζόμαστε σε εσά. έτσι ώστε να προχωρήσουμε δείχνοντας την απαραίτητη φιλοδεξία. Καλή διασυνδεσιμότητα είναι μία από τι ακρογωνίε λίθους για την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων και θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προσφέρουν τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες και τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει ο ψηφιακό κόσμος. Ο κωδικός για τις ηλεκτρονικές ε, συνομιλίες και επαφές είναι ένα βασικό ε, βήμα προς το εμπρός, προς μια κοινωνία του Gigabyte. Και είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες της Εστονικής Προεδρίας. Θα θέλαμε να πετύχουμε συμβιβασμό στο Συμβούλιο για τα θέματα αυτά του κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε και τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Και χαίρομαι που θα συνεργαστώ με την Επιτροπή Ήτρα και είμαι σίγουρη πως θα καταφέρουμε μαζί να προχωρήσουμε προς μια συμφωνία που θα ικανοποιεί όλα τα μέρη για τα θέματα τα ενεργειακά και πιο συγκεκριμένα ε, μαζί με τα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να εξασφαλίσουμε πως θα έχουμε αποτελεσματικό συντονισμό στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επίσης θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε ε, να ε, διατηρήσουμε την βεβαιότητα των επενδύσεων και να λάβουμε υπόψη και τις ιδιάζουσες εθνικές συνθήκες. Πιστεύω πως γενική προσέγγιση θα ε, πετύχουμε και η επόμενη Προεδρία θα προχωρήσει σε τριμερείς διαλόγους. Τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει τη δέσμηση να εξελίξουν δίκτυα 5G. Την επόμενη εβδομάδα θα συζητήσω τι βήματα μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή με τους Υπουργούς Τηλεπικοινωνιών έχουμε ε, εμπλέξει και τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου στη συζήτηση και ελπίζω πως θα στείλουμε ένα στεναρό μήνυμα και θα πούμε χρειάζεται γρήγορα, γρήγορα να ε, αποκτήσουμε αυτό το δίκτυο 5G παντού. Θα πρέπει λοιπόν η ενιαία ψηφία αγορά να θεωρηθεί ως ένα φαινόμενο που εξελίσσεται συνέχεια, που μεταλλάσσεται συνέχεια και να δούμε τι μας περιμένει. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι να καταλήξουμε σε ένα νομικό και πολιτικό πλαίσιο για την οικονομία των δεδομένων δεδομένων. Καταρχήν, είναι αδιαμφισβήτητο ότι να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στα δεδομένα είναι ζωτική σημασία έτσι ώστε η Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια οικονομία. Άρα λοιπόν, για να χρησιμοποιήσουμε στο μέσο αυτά που μπορούν να μα προσφέρουν τα δεδομένα, χρειάζεται να γίνουμε ένωση δεδομένων με σαφεί κανόνε για την ανταλλαγή δεδομένων και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό κλάδο. Άρα λοιπόν η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ελεύθερη ροή ε, των πληροφοριών που αφαιρεί κάποιες ανέτειες, κάποιους ανέτειους περιορισμούς στην κυκλοφορία δεδομένων και ε, στο localization των δεδομένων είναι κάτι πολύ θετικό. Και σίγουρα και εσάς σας φαίνεται πολύ θετική αυτή η εξέλιξη. Όμως αυτό αποτελεί μία μόνο πτυχή της ενδυνάμει ε, ένωσης δεδομένων. Παράλληλα πρέπει να δούμε θέματα που προκύπτουν, όπως για παράδειγμα η πρόσβαση στα δεδομένα και η επαναχρησιμοποίηση των μη προσωπικών δεδομένων. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, εμείς θα κάνουμε μια πολιτική συζήτηση για όλες τις πτυχές της ελεύθερης κυκλοφορίας δεδομένων στο άτυπο που θα κάνουμε τον Ιούλιο στο Τάλιν την επόμενη εβδομάδα και για την αναμενόμενη πρόταση α, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους περιορισμούς των data localization θα κάνουμε μια πολιτική συζήτηση στη συνάντηση του Βουλίου το Δεκέμβριο. Αλλά αυτά είναι μόνο κάποια πρώτα βήματα προς μια ενός δεδομένων και ελπίζω πως το Κοινοβούλιο θα βοηθήσει το θέμα να προχωρήσει και μετά την δική μας Εστονική Προεδρία με τους υπόλοιπους εταίρους μας από το Τρίο Προεδριών. Επίσης, επειδή είχαμε αυτές τις πρόσφατες παγκόσμιες επιθέσεις, είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε. Μία ενιαία ψηφιακή αγορά θα πρέπει να ασφαλιστεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και με τη νέα στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσει ε, μια ε, κυβερνοασφάλεια που θα αποτελεί και βασικό όπλο στη φαρέτρα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και γι' αυτό αναμένουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κυβερνοασφάλεια, την πιστοποίηση και την ε, ετικετοθεσία. Χρειάζεται εμπιστοσύνη, συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ θεσμικών οργάνων. Είναι και αυτό κομβικό σημείο και εμείς θα ξεκινήσουμε τη δουλειά μας για να ανανεώσουμε και να ενημερώσουμε την εντολή της ΕΝΗΣΑ το φθινόπωρο. Να σας πω πως δεν έχω να κάνω μόνο με ψηφιακά θέματα. Εγώ ασχολούμαι και με το διάστημα. Και πρέπει να σας πω πως είναι προτεραιότητα της Εστονικής Προεδρίας να προσφέρει κάτι πραγματικό στην εφαρμογή της σχετικής στρατηγικής στην Ευρώπη. Εμείς δηλαδή θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να υπογραμμίσουμε τις προσπάθειες που γίνονται για να βελτιώσουμε αλλά και να αναδείξουμε την διαστημική πόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να χρησιμοποιηθεί αυτό για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, για να δημιουργηθεί ανάπτυξη, να έρθουν επενδύσεις, να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Δηλαδή έχουμε το εμβληματικό διαστημικό πρόγραμμα που είναι το Κοπέρνικους που αυτή τη στιγμή περνά την ε, ενδιάμεση αξιολόγηση ε, του 14-16. Εμείς θα προετοιμάσουμε συμπεράσματα του Συμβουλίου από τα διδάγματα ε, που έχουμε λάβει από την μέχρι τούδη εφαρμογή του προγράμματος. Αλλά το πιο σημαντικό για το μέλλον του προγράμματος και για την παρατήρηση του πλανήτη γενικότερα. Η άποψή μας είναι να μεγιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα ε, και τα πλεονεκτήματα για τους Ευρωπαίους πολίτες, για την ευρωπαϊκή οικονομία και να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία. Για τον Καλλιλέο, αυτό που έχουμε σκοπό και έχουμε σχεδιάσει είναι να ε, υιοθετήσουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ενδιάμεση αξιολόγηση του κανονισμού GNSS ε, στο σχετικό Συμβούλιο που θα συνδεθεί το Δεκέμβριο. Και ευθυγραμμιζόμενοι με την ψηφιακή ε, ατζέντα της Εστονικής Προεδρίας θέλουμε να τονίσουμε τα πλεονεκτήματα μιας ευρύτερης και ευφιέστερης εφαρμογής της ψηφιακής τεχνολογίας. Θέλουμε να εστιάσουμε στο πώς εμείς κατανοούμε πώς διεκπεραιώνουμε, πώς εκμεταλλευόμαστε τα σχετικά δεδομένα έτσι ώστε αυτά να μεταφερθούν σε καλύτερες, πιο ανταγωνιστικές παγκόσμιες θέσεις εργασίας για τις εταιρείε μας και για καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες στην Ευρώπη. Και ξέρετε πως αυτά θα τα πούμε και στην ε, Ευρωπαϊκή Διαστημική Εβδομάδα του 2017 που θα γίνει στην Εστονία 3 με 9 Νοεμβρίου. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό η ψηφιακή Ευρώπη. Όλοι ξέρουμε πως ο χώρος του διαστήματος είναι, διαστήματος είναι ατέρμονος. Ο ρόλος της Προεδρίας είναι να βρει μια ισορροπία μεταξύ των αντικρουόμενων απόψεων, παραδόσεων και συμφερόντων της Ευρώπης σήμερα και να καταλήξουμε στα καλύτερα δυνατόν αποτελέσματα υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών. Υπογραμμίζοντας λοιπόν τους προαναφερθέντες φακέλους, σκοπεύουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε τους επόμενους 5,5 μήνες που μας μένουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου διαθέσατε χρόνο, που με ακούσατε και είμαι έτοιμη να απαντήσω και στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Εκπρόσωποι πολιτικών ομάδων. Συναδελφοί, παρακαλώ. Δύο λεπτά ο καθένας. Οι άλλοι έχουν δικαίωμα να μιλήσουν ένα λεπτό. Εκτό εκπροσώπων πολιτικών ομάδων. Από το ΕΛΚ, η κυρία Δεκαστή Βέρα. Πρόεδρε, καλώ ήλθατε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ για αυτήν την δυνατότητα ενημέρωση που αποδεικνύουν την που την προσήλωσή σας στην ψηφιακή, στο ψηφιακό θεματολόγιο. σημαντικό μέρος του προγραμματός σας, της Προεδρίας. Η συνδεσιμότητα, επιτρέψτε να πω, είναι η ραχοκοκαλιά της προσπάθειας αυτής. Χωρίς ε, συνδεσιμότητα δεν πρόκειται να μεταμορφώσουμε ψηφιακά την Ευρώπη. Είναι λοιπόν ζωτική σημασία. Κατά τα άλλα, γνωρίζετε καλά ότι ο κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι ένα βήμα στην προσπάθεια βελτίωσης της συνδεσιμότητας. Υπάρχει με την ανάπτυξη δικτύων μεγάλης χωρητικότητας που χρειάζονται σημαντικές επένδυσεις και ούτω καθεξής. Αλλά είναι αυτό που θα ανοίξει το δρόμο και για άλλες συναφείς εξελίξεις. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία μπροστά μας. Υπάρχει δέσμευση. Θα δούμε. Ε, θα συνδυάσουν και οι σκιώδεις εισηγητές και ελπίζω ότι θα εξασφαλίσουμε εν τέλει πολιτική συνένεση. Κατόπιν αυτού, 11 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε και ελπίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με τους τριμερείς διαλόγους. Δεν μπορώ να σας διαβεώσω εσάς ως πρόσωπο του Συμβουλίου, ότι στο τέλος της Προεδρίας σας θα έχουμε πετύχει και πολιτική συμφωνία επί όλων αυτών των θεμάτων. Όμως υποσχόμαστε ότι υπάρχει πολιτική βούληση Βλέπω ότι υπάρχει και η δική σα, αλλά σα πρόσχομαι ότι υπάρχει και η δική μα. Παρακαλώ, από του σοσιαλιστέ Ζωρινιό. Πρόεδρε. Είχα προηγουμένω την ευκαιρία να ευχηθώ κάθε επιτυχία στη συναδελφό σα και ανέφερα και τι μεγάλε προσδοκίε που συνοδεύουν την Προεδρία σα, ειδικά όσον αφορά την Ψηφιακή Ένωση. Η ψηφιακή ένωση είναι βεβαίω πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Αν θέλουμε πραγματικά να οικοδομήσουμε μια ένωση. Ε, μερικά σχόλια επιτρέψτε μου. Πρώτον, πώς θα επωφεληθεί από το Wi-Fi for You, την πρωτοβουλία για δωρεάν διαδίκτυο σε διάφορε περιοχές ανά την Ευρώπη θα το αξιοποιήσετε για να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών, να πιστέψουν στην κοινωνία της πληροφορίας. Πιστεύω ότι θα ήταν καλή ιδέα η Εστονική Προεδρία να αξιοποιήσει ακριβώς τα θέματα ενέργειας μαζί με αυτά της ψηφιακής αγοράς και τα δίκτυα για να τα αναπτύξετε όλα μαζί, να αντιμετωπίσετε το, την ενεργειακή φτώχεια μεταξύ άλλων, να πετύχουμε και τους στόχους του Παρισιού κλπ. Συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους. Και αυτό είναι και το ενδιαφέρον πιστεύω. Γι' αυτό η ευκαιρία είναι ενδιαφέρουσα. Ανοίγει πάρα πολλέ δυνατότητε. Πώ το βλέπετε λοιπόν το θέμα αυτό, Έθεσα το ίδιο ερώτημα στη συναδελφό σα. Το διαδίκτυο είναι ακριβώ αυτό, η συνάντηση των δικτύων. Και αυτά πρέπει να αξιοποιήσουμε. Από την ECR, Καλώ ήλθατε κύριε Υπουργέ. Χαίρομαστε που σας έχουμε εδώ, στην αρχή της Προεδρίας σας. Είπατε, και από το άκουσα, πόσο σημαντικός είναι ο κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο μέλλον. Το είπε και η κυρία Δικαστήγιο. Ε, μία ερώτηση. Ο κώδικας είναι πολύ σημαντικός, ναι, όμως χρειάζεται και κάτι άλλο. Ο Μπερέκ, ο οργανισμός των ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες πρέπει να δημιουργηθεί πραγματικά. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο περισσότερο γι' αυτό. Και η Πιλάρ σε αυτό αναφέρθηκε πρέπει στους δύο αυτούς τομείς να συνδυάσουμε τα θέματα όσο πιο πολύ γίνεται. Η έκθεση δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη στο Συμβουλίο. Θα μπορούσατε εσείς να μας πείτε πώς βλέπετε το θέμα, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και για τον Γαλιλαίο. Αναφερθήκατε στη σημασία της ευρωπαϊκής πολιτικής για το διάστημα και ο το Γαλιλαίο είναι μέρος αυτής της πολιτικής. Είναι μάλλον το μεγαλύτερο έργο στον τομέα, σίγουρα από οικονομική σκοπιά. Θα θέλατε να μας πείτε γιατί περιεκόπη ο σχετικός προϋπολογισμός. Γιατί το ξέρετε ότι περικόπηκε. Εξ ονόματος και άλλων συναδέλφων εδώ πρέπει να πω ότι εξεπλάγημεν όταν ακούσαμε για περικοπές. Γιατί αυτό. Τι συνέβη στο Συμβούλιο. Δυστυχώς έτσι περιπλέκεται η ζωή του έργου. Αυτά. Καλή επιτυχία και πάλι. Δεν θα είναι εύκολο το έργο σας. Δεν είναι πολύ οι έξι μήνες. Θα θυμάστε γιατί έχουμε και το καλοκαίρι. Από την άλλη, και Καλάς. θα αποφελθώ για να ξαναμιλήσω ασθενικά. Λοιπόν, καλησπέρα. Μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά τις δικές αρμοδιότητες. Λέει στην Υπουργό, κύριε Καλάς. Για το service over the top, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό ασθενικά. στο Συμβούλιο μιλήσετε για ηλεκτρονικές επικοινωνίες θα ήθελα να θέσω το εξή ερώτημα. Δεν θα ήθελα να προβούμε σε υπερβολικέ περιτές ρυθμίσεις και να ψηφίσουμε νομοθεσία που δυσκολεύει τα πράγματα. Το θέμα είναι να διευκολύνουμε τις παραδοσιακέ επιχειρήσει. Και μετά μίλησε και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων. Το θέμα του γεωγραφικού εντοπισμού και των γεωγραφικών περιορισμών στην διακίνηση των στοιχείων. Τι θέλουν προκειμένου τα κρατη Θέλουν να προχωρήσουν, το βλέπουν ως καλή ιδέα. Πες μας γι' αυτό. Και τρίτον, τρίτη ερώτηση. Σε σχέση με τον περιορισμό των επικοινωνιών σε περιπτώσεις ε, αντιμετώπισης της τρομοκρατίας κλπ. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα το οποίο ε, προκύπτει κάθε τόσο. Ο κ. Μπουρικόφερ από τους Πράσινους. Πρόεδρε, καλώς ήλθατε κύριε Υπουργέ. τρει ερωτήσει σχέση μεταξύ ψηφιοποίηση και ενέργεια. Το είπαν και άλλοι αυτό βεβαίω. Αλλά πάνω στο ίδιο θέμα. Ένα σχόλιο παρακαλώ όσον αφορά την γενικότερη σχέση μεταξύ ψηφιοποίηση και απόδοση στον ενεργειακό τομέα, στην οικολογία και την κυκλική οικονομία. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά μαζί, γιατί δεν είναι μόνο η ενέργεια, Πώς θα προαγάγετε αυτήν την ε, διασύνδεση, αλληλοσύνδεση, αν θέλετε, αυτών των τομέων και θεμάτων. Δεύτερον, ποια είναι η εκτιμήση ως προς το εξή, Φαίνεται ότι διάφορες διαφορετικές περιοχές στον πλανήτη έχουν εμπλακεί σε έναν αγώνα δρόμου στον τομέα της ψυχικής τεχνολογίας. Πόσο χρόνο έχουμε. Έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου να αποφασίσουμε αν θα κινηθούμε γρήγορα προς το μέλλον ή αν θα χάσουμε αυτόν τον αγώνα δρόμου και θα μείνουμε πίσω. Πού βρισκόμαστε χρονικά. Και τρίτον, το θέμα της αμοιβαιότητας. Σε αυτόν τον αγώνα δρόμου, ξέρετε, υπάρχει και ένας ανταγωνισμός στο θέμα της, ε, των νόμων και των κανονισμών. Ε, δεν ακολουθούν όλες αυτές τις περιοχές του πλανήτη την ίδια προσέγγιση πρέπει να επιμείνουμε στην αμοιβαιότητα, για παράδειγμα, όσον αφορά τον γεωγραφικό εντοπισμό και περιορισμό των δεδομένων. Κάποιες αρχές επιμένουν στον κανόνα. Εμείς δεν είμαστε προφανώς υπέρ. Λοιπόν, τι θα γίνει με το θέμα αυτό. I'm not too fast because... Mm, δεν βιάζομαι γιατί η υπουργό προετοιμάζει τις ε, απαντήσεις της. Είναι δύσκολο να το κάνει κανείς αυτό μέσα σε δύο λεπτά. Περνάμε λοιπόν τώρα στις παρεμβάσεις του ενός λεπτού. Κύριε Κάριντς, όχι δεν θέλετε. Νόμιζα ότι μου ζητήσατε το λόγο. Η κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κυρία Υπουργέ και από μένα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην Προεδρία, στα κάθε κοντά σας και χαίρομαι πολύ που μας παρουσιάσατε ένα τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα. Έχετε την αμέριστη υποστήριξή μου. Δύο θέματα θέλω να ε, θέσω. Ε, ένα στο οποίο δεν αναφερθήκατε, που όμως είναι ε, πολύ σημαντικό για τη χώρα σας και που μπορούν οι άλλες χώρες να μάθουν πολλά από σας. Είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα η οποία να, παρουσιάζει, να προσφέρει τόσες πολλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πολίτες της. Ε, μπορείτε ενδεχομένως να παρουσιάσετε τα επιτεύγματα σας αυτά και στα άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης, ε, δίνοντάς του και το, το, το κίνητρο να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Επίσης, μιλήσατε ε, για την κυβερνοασφάλεια, ότι σκοπεύετε να ενισχύσετε την εντολή που έχετε και ότι θέλετε να καταστήσετε επίκεντρο της Προεδρίας σας και τον τομέα της διαστημικής πολιτικής. Μπορείτε όμως να μας πείτε περισσότερο τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε στον Κοπέρνικο, στον Γαλιλαίο. Ε, αναφερθήκατε στις πρωτοβουλίες και στα προγράμματα αυτά, αλλά τι, τι ακριβώς σκοπεύετε ως συγκεκριμένα και απτά μέτρα να λάβετε ε, στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπον. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Σας εύχομαι. Ελπίζουμε η Ιστονική Προεδρία να ε, δώσει αυτό το νέο, τη νέα πνοή στην ε, ψηφιακή, στο ψηφιακό θεματολόγιο της Ευρώπης. Δύο ερωτήματα. Ποια πιστεύετε ότι είναι η ετοιμότητα των κρατών μελών να, συνεχίσουν, να, να ξεκινήσουν μάλλον τις συζητήσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αλλά και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Και το δεύτερο θέμα επίσης σχετίζεται με την ελεύθερη ε, ροή των δεδομένων αλλά από μια διαφορετική σκόπια. Η εστονική κυβέρνηση παρουσίασε τη διακήρυξή της για την κοινωνία της ψηφιακής υγείας τον Μάρτιο. Είναι κάτι πραγματικά που μας εμπνέει πολύ, κάτι πολύ σημαντικό. Πώς σκοπεύετε να ξεκινήσετε το κοινό, τις κοινέ εργασίες με τα άλλα κράτη-μέλη στο θέμα αυτό και να συνδυάσετε τις προσπάθειες σας ε, με εκείνες της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα παρουσιάσει το φθινόπωρο τη δική της ανακοίνωση σχετικά με την ε, ηλεκτρονική υγεία. Ευχαριστώ. Äh, σα ευχαριστώ πολύ. Έχουμε εξαίρετους ε, διερμηνείς, οπότε θα μιλήσω και εγώ εστονικά. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο, όσου έθεσαν ερωτήματα, υπέβαλαν προτάσεις και παρατηρήσεις. Ελπίζω να μην ξεχάσω τίποτα και να απαντήσω σε όλα όσα ακούστηκαν. Συμφωνώ απόλυτα με την ε, κυρία Καστήλιο. Και είναι λογικό, ακριβώς γιατί έχουμε κοινούς στόχους. Ας ελπίσουμε λοιπόν από κοινού να τους επιτύχουμε. Γενικά, μιλώντας για συνδέσεις, γνωρίζουμε τι σημασία έχει η καλή πρόσβαση στα δεδομένα και στα, στο Wi-Fi. Δεν μπορούμε να μιλούμε καν για ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων αν δεν ε, έχει εξασφαλιστεί η συνδεσιμότητα, η οποία θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, ε, θα πρέπει να καλύπτει όλες τις γεωγραφικές ε, περιοχές ε, αλλά θα πρέπει να είναι και υψηλή ποιότητα από την άποψη ότι τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να μπορούν να ανταλλάσσονται και να κυκλοφορούν γρήγορα και σε μεγάλους όγκους. Ο, για το ερώτημα του κυρίου Σορίνιο σχετικά με, το, με την πρωτοβουλία και το πρόγραμμα Wi-Fi for You. Πρόκειται για μια πολύ θετική πρωτοβουλία, κατά τη γνώμη μας. Περιμένουμε την τελική έγκριση της πρότασης από τους δύο συνομοθέτες και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουμε εντατικές εργασίες ε, τους φθενοπορεινούς μήνες ε, στον τομέα αυτού του προγράμματος του Wi-Fi for You και θα επιδιώξουμε να εξασφαλίσουμε και τη χρηματοδότησή του. Ηλεκτρονικές, ε, ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Πρόκειται για ε, ένα πολύ σημαντικό πακέτο ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν τους υπουργούς και στις 9 ε, Ιουλίου καταλήξαμε σε συμπεράσμα στο Συμβούλιο. Έχουμε λοιπόν πλέον την αναγκαία βάση για να προχωρήσουμε μπροστά. Όσον αφορά δε τον Μπάρακ, τον Μπέρεκ, η προσέγγιση του Συμβουλίου είναι πρώτα να καταρτιστούν τα καθήκοντα, οι στόχοι αυτού και από εκεί και πέρα θα δούμε ποια καθήκοντα, ποιοι τομεί αρμοδιότητας θα προσδιοριστούν ε, μέσω του κανονισμού στο μέλλον. Όσον αφορά το διάστημα, η Εστονία κατά τη διάρκεια, της, ε, κατά τη διάρκεια του ε, Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας του Δεκεμβρίου σκοπεύει να διοργανώσει μια συνεδρίαση όλων των Υπουργών ε, υπεύθυνων για θέματα διαστήματος και στο πλαίσιο αυτό να γίνει μια συζήτηση για την διαστημική στρατηγική η οποία τότε πια θα έχει ε, χρόνο ζωής ενός έτους πια και θα γίνει ένας απολογισμός. Γενικά αυτό που ισχύει είναι ότι για να προχωρήσει ο Κοπέρνικος θα πρέπει να εξασφαλιστούν επιπλέον χρηματοδοτικά μέσα και κονδύλια. Χωρίς κάτι τέτοιο δεν μπορεί να προχωρήσει και θέλουμε πλέον να προσφέρουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και ευρύτερα στις επιχειρήσεις της Ευρώπης να προσφέρουμε και ε, διαστημικά δεδομένα κάθε ε, πολίτης έχει δικαίωμα να ωφελείται από αυτά τα δεδομένα. Η Εστονία μάλιστα έχει πολύ ε, μεγάλη εμπειρία στον τομέα της διαστημικής πολιτικής και έχουμε σκοπό ε, να συμβάλλουμε ε, με, στο, βαθμό των, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας ώστε να διατεθούν αυτού του είδους τα δεδομένα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό είναι ε, σημαντικό, ε, σημαντικό και για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς γιατί μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων, ε, όπως και η ο ψηφιακός εγχρονισμός των κρατών μελών, των διοικήσεων και μέσω της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Δεν υπάρχει και άλλος τρόπος, ε, πρέπει να σας πω. Πρέπει να γίνεται καλύτερη αξιοποίηση και ανάλυση των δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας, προκειμένου να μπορέσουμε να χαράξουμε τα μελλοντικά βήματα. Για το ερώτημα της κυρίας Κάλας. Μια στιγμή να βρω το ερώτημά σας γιατί το κατέγραψα στα χαρτιά μου αλλά δεν μπορώ να το βρω αυτή τη στιγμή. Ανάτο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτο ερώτημα της κυρίας Κάλλας που αφορούσε ε, ε, ενδεχομένως ε, την ε, υπερβολική ρύθμιση ε, των ε, επιχειρήσεων πληροφορικής και επικοινωνιών. Θεωρώ ότι έχουμε ένα πολύ θετικό πλαίσιο και δεν θέλουμε να ε, υπερβάλλουμε στον τομέα αυτόν. Έγιναν συζητήσεις και στην, στον, ε, στο Συμβούλιο και επί Μαλτεζικής Προεδρίας και ε, συμφωνήσαμε όλοι ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες εφόσον είναι παρόμοιες θα πρέπει να διέπονται και από παρόμοιους κανόνες, γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους παίκτε τη αγοράς. Υπάρχει η οδηγία για το περιεχόμενο, το ψηφιακό περιεχόμενο, καθώς και τις άλλες νομικές πράξεις που σχετίζονται με τον ε, τομέα αυτών και σε όλες αυτές τις νομικές πράξεις περιλαμβάνονται οι ίδιες ε, απαιτήσεις για την κρυπτογράφηση. Αυτή τη στιγμή Δεν περιμένουμε ε, προτάσεις ούτε για την κρυπτογράφηση ούτε για τα backdoor, για τα ψηφιακά κενά, για την κυβερνοασφάλεια. Επίσης είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και στο οποίο θα επικεντρωθούμε και στο μέλλον. Την άνοιξη του 2018 θα έχουν πλέον βάσει του χρονοδιαγράμματος τεθεί σε ισχύ όλες οι σχετικές οδηγίες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποσχεθεί ότι θα υποβάλει έως το Σεπτέμβριο μια νέα στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια. Η στρατηγική που ισχύει σήμερα ε, είναι 4-5 ετών. Δεν είναι και ακριβώς παλιά. Παρ' όλα αυτά οι εξελίξεις στον ψηφιακό κόσμο είναι ε, πολύ πιο ε, γρήγορες Γι' αυτό και την ε, έχουν καταστήσει εν μέρη τουλάχιστον παροχημένη. Χρειάζεται λοιπόν να επικαιροποιήσουμε και εμείς την δική μας στρατηγική, να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας και να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή των ε, οδηγιών μας. Στην τελευταία ε, κυβερνοεπίθεση που έγινε, οι εταιρείες που επλήγησαν ήταν όλες διεθνείς επιχειρήσεις. Γι' αυτό και είναι σημαντικό η κυβερνοασφάλεια. Βεβαίω δεν αρκεί να είναι υψηλή η κυβερνοασφάλεια στην Εστονία, στην Εστονία αλλά στι άλλε χώρε να μην είναι υψηλή. Χρειάζεται εναρμόνιση. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Πράγματι στην Εστονία έχουμε επιτύχει πολλά. Έχουμε επικεντρωθεί σοβαρά ε, ως προς την πρόοδό μας ε, στον τομέα αυτό και τον Νοέμβριο αν δεν κάνω λάθος, θα διοργανώσουμε και μια συνδιάσκεψη υψηλού επίπεδου σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπου και θα εγκριθεί μια, διακυβέρνηση, μια διακήρυξη για το ποια θα, μπορούσαν να είναι τα, ποια θα πρέπει να είναι τα μελλοντικά ε, μέτρα και πώς θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε την ε, ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη Ιδίω δε την εφαρμογή της αρχής κάθε έγγραφο να ζητείτε, να υποβάλλετε αίτηση για κάθε έγγραφο μία φορά και σε ένα μόνο σημείο. Τελευταίο ερώτημα που αφορούσε τον Γαλιλαίο. Για τον προπολογισμό αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα, περνά, ότι θα κάνουμε ό,τι περνά από το, χέρι, μας. Ακόμη και αν λοιπόν μειωθεί ο προπολογισμό, θα εξασφαλίσουμε να επιτευχθούν ε, να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή πρόοδος. Ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων επίσης ήταν ένα θέμα που έθεσαν πολλοί ε, ευρωβουλευτές, πολλά μέλη, πολλά της Επιτροπής σας. Σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε το έργο μας επί του θέματος αυτού. Περιμένουμε και τη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν. Το Σεπτέμβριο δε διοργανώνουμε και μια πολιτική συζήτηση για το θέμα αυτό. Ελπίζω λοιπόν να απάντησα σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν. Είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας. Ελπίζω να σας δω και στην Εσθονία, όπου και διοργανώνουμε 50 διαφορετικές ε, διασκέψεις για ζητήματα που άπτονται του, της ψηφιακής οικονομίας και του ψηφιακού κόσμου. Ακριβώς γιατί για εμάς στην Εστονία αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό δεν, ε, δεν θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο κάποιους ειδικού, κάποιους εμπειρογνώμονες. Είναι ένα θέμα που αφορά όλο το, το, όλους τους υπουργούς και φυσικά με τη δική σας συμμετοχή θα καταφέρουμε να επιτύχουμε ακόμα περισσότερα. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω πως ε, Κάνατε μια προσπάθεια, δεν είναι βέβαια δυνατόν να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με λεπτομέρειες, αλλά ξέρουμε πως κάτι τέτοιο είναι αδύνατον. Οπότε, είναι πολύ σύντομη η συνάντησή μας και για να καταφέρουμε να απαντήσουμε σε όλους τους συναδέρφους, ίσως θα έπρεπε να πάρετε ένα κατάλογο ερωτήσεων πίσω μαζί σας στο Τάλιν και αν έχετε κάτι να μας το στείλετε σε απάντηση έτσι ώστε να ανταποκριθείτε και στις δικές μας προσδοκίες. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ κυρία μου για την παρουσίαση που κάνατε και επίσης για όλες τις απαντήσεις που μας δώσατε. Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία για το επόμενο εξάμεινο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για μένα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ήταν ωραίες οι ερωτήσεις, ήταν καλά τα σχόλια και ελπίζω να τα πούμε στο Τάλιν. Ξέρω πως σύντομα ξεκινάτε τις θερινές διακοπές, οπότε σας εύχομαι και καλό καλοκαίρι. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αυτό που συμβαίνει πάντοτε στις συναντήσεις μας. Δηλαδή, Νομίζω ότι ανταποκρίνομαι στα όσα πιστεύει ο κύριος Ράινχολτ. Συμβαίνει πάντα. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε με λεπτομέρειες σε όλα. Όμως έχουν καταγραφεί ερωτήσεις, ερωτήσει, θα συνοδεύσουν τις προσκεκλημένες μας, οπότε σας παρακαλώ πολύ και εσείς να θυμηθείτε τι ρωτήσατε έτσι ώστε ε, να σας απαντήσουν. Δεν έχω τίποτα εναντίον των ερωτήσεων που κάνατε. Είναι πάρα πολύ λογικές και είναι εξαιρετικό που κάνουμε τόσο λεπτομερείς ερωτήσεις. Και νομίζω ότι σίγουρα δεν θα έπρεπε να τις αποφεύγουμε, αλλά δεν είναι δυνατόν να τα απαντάμε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση που θέλετε να κάνετε, όσο λεπτομερείς όσο λεπτομερείς και αν είναι ερώτηση αυτή, μην διστάσετε, έχετε κάθε δικαίωμα να την κάνετε. Θα δώσω τώρα το λόγο τώρα στην κυρία Μαΐλης Ρέψ, που είναι η Υπουργό Παιδείας και Έρευνας. Το θέμα μας λοιπόν. Έρευνα. Έρευνα και διάστημα. Και εξ όσων γνωρίζω, η κυρία Ρέψ δεν είναι υπεύθυνη μεν για την καινοτομία, αλλά για μας τα θέματα αυτά συνδέονται τόσο πολύ έρευνα, καινοτομία, που θα ήθελα να μην σας προξενήσει έκπληξη κυρία μου, αν σας κάνω και κάποιες ερωτήσεις για θέματα καινοτομία. γιατί δεν μπορούμε εμείς να τα αφαιρέσουμε από το θέμα αυτό τόσο αστηρά και αν χρειαστεί μπορείτε να μεταφέρετε τις ερωτήσεις αυτές σε οποιονδήποτε άλλο υπουργό στη δική σας κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να δούμε τα θέματα παιδείας, θέλουμε να δούμε τα θέματα έρευνας, καινοτομία. Είναι δηλαδή το τρίγωνο της γνώσης, που είναι πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει αυτό το τρίγωνο να διατηρηθεί ως έχει. Και να μην αφήσουμε ε, οτιδήποτε απ' έξω. Θα μιλήσουμε και για το Horizon 2020, για το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο και βέβαια στην παιδεία, εμείς δεν είμαστε Επιτροπή Παιδείας, αλλά έρευνα παιδεία είναι δύο αλληλένδετα θέματα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ αξιότιμη κύριε Μπούζα και ήταν πραγματικά καταπληκτικό που συναντηθήκαμε και για λίγο προηγουμένως και σίγουρα θα τα πούμε πολύ συχνά, είμαι σίγουρη τους επόμενους μήνες. Αγαπητοί συνάδελφοι του Κοινοβουλίου, είναι για μένα πολύ μεγάλη χαρά να βρεθώ σήμερα κοντά σας και να έχω αυτή την πρώτη πολύ σύντομη επαφή και ανταλλαγή απόψεων για τις προτεραιότητες μας, μια και τώρα έχουμε την Προεδρία του Συμβουλίου. Και Παράλληλα, θα πάρω μαζί μου τις δικές σας ιδέες, αυτά που είπατε σήμερα, μέσω των πιο άτυπων επαφών που κάναμε σήμερα με διάφορα μέλη, γιατί ήταν όλα πάρα πολύ ενημερωτικά και θα ήθελα επίσης να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω από των προτέρων, γιατί όλα τα θέματα και οι συζητήσεις που έχουν γίνει εδώ και για το Horizon 2020 και για άλλες προτεραιότητες δικής μας προεδρίας. Τα έχουμε παρακολουθήσει στενά. Είναι η πρώτη φορά που η Ιστονία αναλαμβάνει η προεδρία. Ήμασταν πάντα η χώρα που ο πληθυσμός στηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε για μας είναι και πιο εύκολο να έχουμε αυτή την ενωμένη προσέγγιση και αυτή την ενωμένη κατανόηση για το τι θα είναι το καλύτερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό και στο χώρο της έρευνας γιατί θέλουμε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε και να δώσουμε μια προστιθέμενη αξία μέσω της έρευνας σε όλους μας. Θα μιλήσω για κάποιες από τις προτεραιότητές μας, θα ήθελα να τονίσω πως με χαρά θα κάνω και άλλες συζητήσεις μαζί σας και με μεγάλη χαρά θα ακούσω σχόλια από εσάς. Αυτή τη στιγμή η Εστονική Προεδρία διανύει μία εποχή που συζητάμε το τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020 και έχουν και κάποια υπαρξιακά ερωτήματα για το μέλλον της ίδιας Ευρώπης. Και πολλές από τις δράσεις που έχουμε αναλάβει εστιάζουν στο να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Η ευρύτερη πολιτική μας στόχευση έχει να κάνει με τη μείωση της απεσιοδοξίας. Ένα ανάχωμα στην απεσιοδοξία έτσι ώστε ε, να τα πάμε καλύτερα στην Ευρώπη και σίγουρα ε, ο χώρος της έρευνας και της καινοτομίας και η συνεργασία εκεί είναι ένας από τους πιο αισιόδοξου και θα δούμε τι θα γίνει με το Horizon 2020 και πρέπει να σας πω πως το τρέχον πρόγραμμα πλαίσιο έχει ακόμα τρία χρόνια για να τρέξει αλλά γίνονται συζητές για το, συζητήσεις για το μελλοντικό πρόγραμμα και γίνεται και η συζήτηση εδώ σε εσά έχουμε και την έκθεση Λαμή και έχουμε τα όσα συζητάνε οι εμπλεκόμενοι. Θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ το Κοινοβούλιο για τη σφαιρική έκθεση που κάνατε για την ενδιάμεση αξιολόγηση και εξέλιξη του Χωράζων 2020. Ήταν η πρώτη τέτοιου είδους και ήταν πάρα πολύ σφαιρική για το μέλλον για το μελλοντικό πρόγραμμα πλαίσιο, νομίζω ότι έχουμε μια κοινή κατανόηση πως υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει να αποφασίσουμε και να σπρώξουμε ως προτεραιότητες κατά την Προεδρία μας. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τη χαρά να πάμε σε μια διάσκεψη με πολλούς από τους συναδέλφους σας και με τη Σολεδάδ Καβεσόν, όπου σε ένα πάνελ που Καθίζαμε μαζί, ξεκινήσαμε μια συζήτηση για το πώς θα είναι το πρόγραμμα μετά το 2020. Είπαμε, συνεργασία, συνεργασία και σε θέματα καινοτομία και είναι πολύ φανερό πως δεν υπάρχει έρευνα χωρίς καινοτομία και το αντίστροφο. Είναι πολύ στενά συνδεδεμένο, οπότε θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις και τι λέει η έκθεση Λαμή σχετικά. Γιατί εδώ υπάρχει το εξή ε, που προκύπτει. Δεν υπάρχει έρευνα χωρίς παιδεία. Κάτι το οποίο καμιά φορά ξεχνάμε, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση στιάζει περισσότερο στο ένα θέμα παρά στο άλλο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε αριστεία και για να πετύχουμε την αριστεία αυτή πρέπει να βασιστούμε σε μια πολύ γερή παιδεία. Και αυτά θα συζητηθούν και σήμερα. Επίσης, Συζητώντας το μέλλον του ευρωπαϊκού προπολογισμού, νομίζω ότι θα πρέπει να μπορούμε να παρουσιάσουμε καλύτερα επιχειρήματα, γιατί πρέπει να επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην έρευνα και στην καινοτομία. Γιατί πρέπει να επενδύσει πιο πολύ από ό,τι μέχρι σήμερα. Και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν πως το κομμάτι αυτό της έρευνας και της τεχνολογίας έχει πολύ θετικές επιπτώσεις για την κοινωνία και για την ανάπτυξη. Και νομίζω ότι αυτό το έχουμε τοποθετήσει προς το προτεραιότητα της Προεδρία μας. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι αυτή τη γνώση να την μεταφέρουμε και να την έχουμε ως πιστικά επιχειρήματα για όσους θέλουν μείωση στον προπολογισμό και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να έχουμε ένα καλύτερο αφήγημα για το τι σημαίνει η έρευνα για την Ευρώπη. Είμαστε πολύ περήφανοι για την ηλεκτρονική Εστονία, το e-Estonia στη χώρα μας, αλλά η επιτυχία αυτού του προγράμματος δεν θα ήταν δυνατή χωρίς καλή βασική έρευνα. Είναι μια μακρά διαδικασία όπου η νέα γνώση, όπου η καινοτομία έχουν αποτελέσει τα βασικά θεμέλια για τις επιτυχίες μας και είναι ένα από τα μεγάλα παραδείγματα ε, της τεράστιας αλλά δύσκολο να ε, υπολογιστεί ε, συνέπειες που έχει η ακαδημαϊκή έρευνα στην οικονομία τη Εστονία. Τα είπα άλλωστε και με τον Πασκάλ Λαμί την περασμένη εβδομάδα, όπου μιλήσαμε για τη χρηματοδότηση. Δεν θέλουμε απλώ να κάνουμε του καλού στην επιστήμη. Όχι. Με τον τρόπο αυτό διατηρούμε και την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Χρειαζόμαστε την καινοτομία, την έρευνα για να ανταποκριθούμε στι προκλήσει του μέλλοντο και να έχουμε κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα. Είναι η έρευνα και η, η καινοτομία αυτέ οι οποίε θα μα. Ε, δώσουν πνοή, θα μας εμπνεύσουν. Και θα πρέπει να έχουμε μία από την βάση προς την κοροφή προσπάθεια να έχουμε περισσότερη έρευνα στην Ευρώπη. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτή είναι η λυπηρή αλήθεια, είναι κάτω από το στόχο του 3% σε επενδύσεις στην έρευνα και αντί το 3% είμαστε στο 2,03% το 2015. Το 90% της δημόσιας επένδυσης σε ε, τεχνολογία και έρευνα είναι σε εθνικό επίπεδο, μόνο 10% σε ευρωπαϊκό και γι' αυτό στην Προεδρία μας δεν θα ασχοληθούμε μόνο με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό αλλά και με τις εθνικές προσπάθειες για να αυξηθούν οι επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία. Όταν μιλάμε για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο, θα πρέπει τότε το Συμβούλιο να στείλει ένα στεναρό μήνυμα. Πώς θα εξασφαλίσουμε πως το πρόγραμμα αυτό θα έχει πολλές επιπτώσεις. Δηλαδή, έχουμε την συνεισφορά των εμπλεκόμενων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη έκθεση Ισλαμή και αυτά αποτελούν τη βάση για τη συζήτησή μα. Είναι η προτεραιότητα. Και εμεί θέλουμε να εξορθολογήσουμε ε, την χρηματοδότηση ε, ευρύτερα στην έρευνα και στην κοινοτομία στην Ευρώπη. Είναι αρκετά ε, περίπλοκο και εμείς θέλουμε να αυξήσουμε τη συνεκτικότητα και την διαφάνεια των εταιρικών συμφώνων στην έρευνα και την ε, καινοτομία, γιατί είναι πολύ περίπλοκη η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και αυτό είναι ένα θέμα που επαναλαμβάνεται ακόμα και στο πλαίσιο του Horizon 2020. Γιατί, γιατί έχουμε όλο και μεγαλύτερο αριθμό ε, εργαλείων, πρωτοβουλειών που αποτελούν το 25% του συνολικού προϋπολογισμού για το Horizon 2020. Και αυτό το μερίδιο σε κάποιο κομμάτι του Horizon 2020 έχει, είναι συνέχεια, δεν είναι αυξανόμενο και έχει φτάσει το 60% όπως λέει και η έκθεση Λαμή, ο ελάχιστο ο στόχος θα πρέπει είναι να καταργήσουμε το 1 τρίτο των ε, χρηματοδοτικών σχεδίων, ε, των εργαλείων και των ακρονίμων. Και αυτό ε, για να έχουμε μια καλύτερη και πιο στρατηγική προσέγγιση στις εταιρικές σχέσεις, στην έρευνα και την κοινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη συνεκτικότητα και να είμαστε ανοιχτοί στους νέους, στους νέους ερχόμενους. Άρα λοιπόν θα σχεδιάσουμε κάποια συμπεράσματα του Συμβουλίου για την αξιολόγηση, την ενδιάμεση του του 2020 για τις μελλοντικές προσεγγίσεις ε, στα προγράμματα πλαίσιο. Επίσης, σας καλώ ελάτε σε μία διάσκεψη για την Ευρωπαϊκή Άριστη Έρευνα Επίπτωση και Αξία για την Κοινωνία. 12 Οκτωβρίου στο Τάλιν. Με υψηλού επίπεδου συζήτηση για να αυξήσουμε και να μεγιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις και την αξία της έρευνα, έτσι ώστε να βρούμε νέα επιχειρήματα για να αυξήσουμε τι επενδύσει σε τεχνολογία και έρευνα στην Ευρώπη. Επιτρέψτε μου να κλείσω λέγοντας πως αυτή η Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συνεργασία μεταξύ των θεσμών, των θεσμικών εργάνων, με τους ερευνητέ, τα Ινστιτούτα που προσφέρουν γνώση και τον βιομηχανικό κλάδο είναι ζωτική σημασία για να έχουμε και να πετύχουμε ένα ε, φιλόδοξο όραμα για την έρευνα και την κοινοτομία στην Ευρώπη μετά το 2020. Ευχαριστώ πολύ. όλα πολύ σημαντικά από το ΕΛΚ. Καλώ ήλθατε κύριε Υπουργέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάτε μεγάλη προετοιμασία, το αντιλαμβανόμαστε και ήταν ενδιαφέρον το πόσο μικρές χώρες προετοιμάσουν τόσο καλά την Προεδρία του ιδιαίτερα στον τομέα τη Έρευνα. Δεν συμβαίνει πάντοτε αυτό και καμιά φορά δεν συμβαίνει ούτε με μεγάλα κρατημέλη. Ε, μια ευθεία ερώτηση. Η απόφαση για τον προπολογισμό, όπω ξέρετε, αναμένεται και έχει σχέση με την έκθεση Λαμή, του λόγους που ακούσαμε την Κυριακή. Αλλά τι γίνεται τώρα Νομίζω ότι έχουμε αποτύχει παταγωδό όσον αφορά τον στόχο του 3% το 2020. Και είπατε ότι είναι ο ενωσιακό προπολογισμό είναι πολύ μικρό έχει περικοπεί και άλλο σε σχέση με του παλιού μα στόχου για το 2020 σημαίνει λιγότερε δαπάνε για τη βιομηχανία που για μένα αυτό είναι το ανησυχητικό. Εν πάση περιπτώσει Εν τέλει, το θέμα είναι τα λεφτά. Και το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό η Προεδρία σα θα υποστηρίξει την φιλοδοξία του Κοινοβουλίου στον προπολισμό. Δηλαδή, για 120 δισεκατομμύρια είναι μια πολύ φιλοδοξή πρόταση με την έννοια ότι η έκθεση Λαμή ε, λέει ότι για να φτάσουμε τα 300 δις πρέπει να αυξάνουμε τα τις δαπάνες μας 150 δις το χρόνο. Αλλά κοιτάξτε τι γίνεται στην Ασία, στην Βόρεια Αμερική, τελείως διαφορετικές αγορές. Και θα το δούμε και στην Κίνα και σε άλλες χώρες της Ασίας. Οι Αμερικανοί τι έκαναν, αύξαναν τον προϋπολογισμό τους, ενώ εμεί ε, τον μειώνουμε. Το περιγράψετε λίγο ουδέτερα, αλλά θα υποστηρίξετε μια πιο φιλόδοξη πρόταση για τον προπολογισμό, η οποία θα μπορούσε να ε, προέλθει και από την Κομισιόν. Και πρακτικά έχουμε ένα πρόγραμμα αριστείας μπροστά μας όσον αφορά την κοινοτομία, αλλά ακόμη ακολουθούμε τους άλλους. Από το Σεπτέμβριο του 2013 Έχουμε διάφορες προσδοκίες. Θα βοηθήσει η Προεδρία σας να κλειστώ το χάσμα, γιατί προχωράμε πολύ αργά, υπερβολικά αργά. Εσείς ενστερνίζεστε την αρχή της αριστείας. Θα ήθελα να ακούσω κάτι πρακτικό από την πλευρά σας, αν θα μας βοηθήσετε. Πρόεδρος, και τώρα, κυρία Βομπάτσικα, εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τι χαρά να ξαναβλέπω την Υπουργό. Ήδη τα είπαμε το πρωί, μιλήσαμε για εκπαίδευση. Σήμερα όμως μιλάμε μόνο για, απόψε μάλλον, μιλάμε μόνο για έρευνα. Τρεις ερωτήσεις. Πώς βλέπετε το εξής θέμα και, και συνεφώς τι δράση θα αναλάβετε όσον αφορά το τρίτο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα για να μειώστε τις περιφερειακές αδικίες, ανισότητες. Πάνω από το 60% των κονδυλίων, όσο αυτή τη στιγμή, έχουν απορροφηθεί σε τέσσερις χώρες και αυτό αποτελεί τεράστιο πρόβλημα. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Τελευταία πήγαμε μόνο σε τέσσερις χώρες. Είπατε εταιρική σχέση, συνεργασία, ναι, αλλά εδώ θα ήθελα να δω αυτήν τη συνεργασία. Τι σκοπεύετε να κάνετε. Άλλο ερώτημα. Θα υποστηρίξετε την πρόταση του Κοινοβουλίου να υποστηρίξει το θεσμό της αριστείας στα διπλώματα βρισιτεχνίας για να μην χαθούν έργα τα οποία έφυγαν και πέταξαν επειδή δεν υπήρχαν αρκετά κονδύλια. Και τρίτον, ενώ και που είπε ο προηγούμενος ομιλητή. Δεν θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε συνεργεία μεταξύ έρευνας και των τεράστιων κονδυλίων που δαπανούμε για την άμυνα. Γιατί να μην δέσουμε το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα με την άμυνα. Δυστυχώς εκεί δεν βλέπω καμία πρόοδο σε αυτές τις μηχανές τρομές, μηχανές που κατάλληλα προκαλούν το θάνατο. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Κύριε Στουσονόσκι από την ομάδα ECR. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας καλωσορίσω και εγώ από την πλευρά μου. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ μαζί μας και είναι ευπρόσδεκτα τα όσα μας είπατε σχετικά με την έρευνα. Η έρευνα είναι η συμβολή μας για το μέλλον. Ενός μέλλοντος το οποίο μάλιστα εμείς μπορεί και να μην ζήσουμε να το δούμε. Είναι σε κάθε περίπτωση σημαντικό να, να συζητήσουμε το θέμα του Horizon 2020 και του Brexit και μάλιστα να τα δούμε από κοινού. Γνωρίζετε ότι η Μεγάλη Βρετανία ήταν ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες της πανεπιστημιακής έρευνας. Τώρα πια το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 ε, οδεύει προς το τέλος του, το 2020 και πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει, όχι μόνο από την άποψη του Brexit, αλλά ιδίως ως προς την συμβολή της Βρετανίας ε, στην ε, έρευνα και ανάπτυξη. Πώς θα προετοιμαστούμε εν ώψη λοιπόν της αποχώρησης Βρετανίας. Ξέρω ότι οι σχετικές διαπραγματεύσεις δεν έχουν αγγίξει ακόμη το θέμα της έρευνας. Όμως νομίζω ότι πρέπει να το κάνουν σύντομα. Διότι πιστεύω ότι στο τέλος θα καταλήξουμε σε ένα φιλικό διαζύγιο. Ελπίζω λοιπόν οι σχέσεις μεταξύ των πανεπιστημίων μας να παραμείνουν ε, ανέπαφες από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου διότι το Ηνωμένο Βασίλειο ε, είναι ηγέτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην πανεπιστημιακή έρευνα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για τα όσα μας είπατε κατά τα άλλα. Ευχαριστώ η κυρία Κάλας από, την, ε, από τους φιλολευθέρους και την Εστονία που ίσως είναι και το βασικότερο χαρακτηριστικό σας σήμερα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναθέσω βεβαίως τα ερωτήματά μας στα εστονικά. Δύο είναι τα ερωτήματα που θέλω να θέσω. Υπάρχουν πολλά καλά προγράμματα για τη χρηματοδότηση της επιστήμης και της έρευνας. Αυτό όμως που λείπει είναι η διασύνδεση των διαφόρων αυτών προγραμμάτων. Το κάθε πρόγραμμα έχει μια αυτόνομη δική του ε, εξέλιξη και πορεία. Το ερώτημά μου προς εσάς λοιπόν είναι ε, σχετίζεται μάλλον και με το τελευταίο ερώτημα που σας θέθηκε. Έχει η Εστονική Προεδρία κάποιο σχέδιο, κάποιο πρόγραμμα προκειμένου να ενισχυθούν οι συμπράξεις, οι συνέργειες. Δεύτερο ερώτημά μου αφορά τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη. Σκοπεύει η Εστονία να αναλύσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί για την ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη. Ο κύριος Τούμες από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. Υπάρχει μια έννοια στα αγγλικά ε, που ε, είναι το white elephants δισεκατομμύρια. Όταν λοιπόν μιλούμε για ένα πρόγραμμα, μιλούμε για έναν ε, αντιδραστήρα στην πραγματικότητα, για μια σύνδεξη πυρηνική, ε, η οποία μπορεί να προκαλέσει, να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Δηλαδή έχουμε αφενός τις περικοπές του προπολογισμού, δύο προγράμματα σύνδεξης και κανείς δεν έχει ε, αναφερθεί σε αυτά. Ε, μιλάμε δηλαδή πραγματικά για την αξία των δαπανών και πρέπει κάποιος επιτέλους να πει είχαμε μεγάλες ελπίδες ε, από αυτά τα προγράμματα και τελικά ε, μάλλον πήγαν στο βρόντο. Ε, δεν πρέπει να γίνει αυτό. Πρόκειται για 2.000 εξαιρετικά μυαλά που ε, εργάζονται σε αυτό τον τομέα και πρέπει να αξιοποιηθούν. Δεύτερον, βιομηχανική πολιτική και καινοτομία. η Κίνα είναι ένας πολύ καλός παίκτη. Ολοκλήρωσε την ε, βιομηχανική της στρατηγική για την ηλική ενέργεια. Εμείς μάλλον από την άλλη πλευρά ε, δεν ε, χρειάστηκε μάλλον να περάσουν 3-4 χρόνια. Γιατί, γιατί δεν μπορούσαμε να βρούμε μισό δις ή ένα δις τέλο πάντων προκειμένου να αξιοποιήσουμε τους πόρους και τους καλύτερους εγκεφάλους και τα καλύτερα εργαστήρια που παράγουν την πιο προηγμένη τεχνολογία σε ολόκληρο τον κόσμο ε, και γιατί ε, διότι δεν είμαστε σε θέση να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ ε, έρευνας και βιομηχανίας. Το ίδιο ισχύει για τη χωρητικότητα των μπαταριών έχουν καταβληθεί ε, μεγάλες προσπάθειες. Αν δεν καταβάλουμε όμως μεγαλύτερες θα χάσουμε από την Ασία. Εγώ είμαι αισιόδοξο άνθρωπος γενικά. Κάθε πρωί ξεκινάω τη μέρα μου με χαμόγελο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ε, εντοπίσουμε βεβαίως και τις αδυναμίες μας και να ε, αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο αυτούς τους ε, λευκούς ελέφαντες, τα white elephants όπως σας είπα στην αρχή. Ευχαριστώ συνάδελφε. First of all, um, uh, members of um, European Parliament, it's. Um, Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά που διαπιστώνω ότι έχουμε μια συναντήληψη στα βασικά ζητήματα. Μας ανησυχεί και μας ε, το θέμα που ανέφερε ο κύριος Τούρμες. Το γεγονός δηλαδή ότι η Ασία και όχι μόνο η Κίνα, είναι και η Ινδία, είναι και η Κορέα, ε, σημειώνει πολύ μεγάλη και πολύ γρήγορη πρόοδο. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τον πιο παραδοσιακό μας ανταγωνιστή, της ΕΠΑ. Κάνουμε συζητήσεις ε, και ε, ρεαλιστικά ε, πρέπει να σας πω ότι εξακολουθούμε να είμαστε 28 κράτη-μέλη, όχι 27 ακόμη. Και υπάρχουν βεβαίως διαφορετικές απόψεις, διαφορετικά συμφέροντα. Έχουμε ωστόσο ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Έχουμε τους ερευνητές μας, έχουμε τα εργαστήρια, έχουμε ένα ελεύθερο ε, ερευνητικό και ακαδημαϊκό πλαίσιο ε, το οποίο εξασφαλίζει την αυτονομία και την ελευθερία της έρευνας και ε, να μην το ξεχνάμε αυτό. Το, το πλεονέκτημά μας είναι το γεγονός ότι κάθε ερευνητής είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Δεν ε, του επιβάλλουμε εμείς κατευθυντήριες γραμμές. Μπορούν να κάνουν μάλιστα μακροπρόθεσμα πολύ σημαντικά πράγματα. Ταυτόχρονα όμως βεβαίως θέλουμε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ έρευνας και καινοτομίας ε, και περισσότερες συμπράξεις. Και αυτό είναι και μια από τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Δύο συγκεκριμένα ε, στόχους έχουμε θέσει. Να εξορθολογήσουμε αφενός ε, την χρήση των πόρων, όπως είπε και η κυρία Λομπάτσκα, γιατί πράγματι είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι πράγματι είμαστε σε θέση να ελιχθούμε σε αυτόν τον ωκεανό. Ε, διότι υπάρχουν διάφορα προγράμματα, υπάρχουν διάφορες εταιρικέ σχέσεις, διάφορες συμπράξεις. Πρώτα λοιπόν πρέπει να ξεκαθαριστεί το τοπίο και να δούμε πού μπορεί να υπάρξει ε, εξορθολογισμός. Ένα τρίτο είναι υπερβολικά φιλόδοξο στόχο, όπω είπατε κι εσεί, παρόλα αυτά θα τον επιδιώξουμε. Δεύτερο ζήτημα που σχετίζεται με την ε, ανταγωνιστικότητά μα, ε, άπτεται και των προτάσεων του Κοινοβουλίου και τη Έκθεση Λαμή. Να υπάρξει σημαντικά υψηλότερη χρηματοδότηση σε εθνικό αλλά και σε ενωσιακό επίπεδο. Σχετίζεται αυτό το θέμα και με το επίπεδο των φιλοδοξιών μας. Στο Συμβούλιο έχουμε ξεκινήσει τις σχετικές συζητήσεις, αλλά βεβαίως κάθε αρμόδιος για την έρευνα συμφωνεί ότι χρειάζεται να επιδείξουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία. Το πρόβλημα είναι βεβαίως ότι χρειάζεται και να πάμε λίγο παραπέρα την συζήτηση αυτή και να καταδείξουμε πώς με απτούς τρόπους η έρευνα και η καινοτομία ωφελεί την οικονομία. Και πολλές φορές αυτό ε, ε, ε γίνεται φανερό και σε συζητήσεις που έχουμε με πανεπιστημιακούς, με ερευνητές. Τώρα λοιπόν προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή και με τους Ευρωπαίους νομοθέτες και με τους εθνικούς νομοθέτες για να τους αποδείξουμε και να τους πείσουμε για το πόσο η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να ωφελήσουν την οικονομία. Τώρα, για τη συγκεκριμένη πρόταση, αν θα είναι 120 ή και διπλάσια ακόμη, εδώ βεβαίως πρέπει να σας πω ότι βασιζόμαστε σε εσά. Διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε ήταν πολύ σημαντικός ε, φορέας για την ενίσχυση ε, των προγραμμάτων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο, ε, αλλά έχουμε ε, σαφώς καθορίσει ότι η πρόταση που θέλουμε να υποβάλει η Κομισιόν θα πρέπει να είναι φιλόδοξη. Για το ερώτημα του κ. Τζανόφσκι και το Brexit. Φυσικά μας απασχολεί και μας πάρα πολύ αυτό το ζήτημα. Βρισκόμαστε σε πολύ αρχική ε, φάση βεβαίω των παραπραγματεύσεων. Δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθούν οι διαπραγματεύσει αυτές στο τέλος, αλλά όσον αφορά την έρευνα, αλλά και για τους άλλους τομεί αρμοδιότητά σας, ε, αν δείτε τους νέους ανθρώπους, καθηγητέ, ερευνητέ, φοιτητέ, όλοι ανησυχούν, και στη Βρετανία δηλαδή. Γιατί ε, είναι σαφές ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην χαθεί αυτή, αυτό το πλεονέκτημα αυτής της ε, αμοιβαίας εποφελούς σχέσης και των ε, προγραμμάτων ε, κινητικότητας μέσω των οποίων μπορούν να συνεργάζονται πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Φυσικά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πού βρισκόμαστε σε αυτό το τομέα, αλλά εφόσον όλες οι πλευρές έχουν κοινούς στόχους, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην μπορέσουμε να βρούμε μια ε, θετική λύση στο θέμα αυτό. Όσον αφορά ε, τη μελλοντική χρωματοδότηση των προγραμμάτων, νομίζω ότι η αφετηρία που έχουμε ε, αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλή. Έχουμε καλά επιχειρήματα, έχουμε ενδιάμεσες εκθέσεις πάνω στις οποίες μπορούμε να βασιστούμε και έχουμε και προτάσεις βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι πράγματι ανταποκριθήκαμε στις υποχρεώσεις μας. Έχουμε ε, ε, στόχους ε, για το πώς μπορούν να ενισχυθούν οι συμπράξεις, πώς μπορεί να ωφεληθεί η οικονομία και για το πώς μπορούν να διασυνδεθούν καλύτερα τα διάφορα προγράμματα. Αν μάλιστα εξετάσουμε και πρωτοβουλίες όπως είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, ή διάφορες συνέργειες ή την πρόταση για τα διαρθρωτικά ταμεία για το πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν διαρθρωτικά ταμεία ή και άλλα ταμεία ε, για την πρόθεση της έρευνας ε, θα δείτε ότι αυτές οι συμπράξεις μπορούν ε, να αποφέρουν περισσότερη χρηματοδότηση και, στην, και για την έρευνα. Ξέρετε ότι υπάρχουν και προτάσεις ώστε και τα αγροτικά ε, ταμεία θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν ε, την έρευνα. Το ίδιο ε, ισχύει και για τις αμυντικές δαπάνες, όπου έχουμε επίσης παρόμοια στάση. για την αριστεία. Από την εστονική εμπειρία ε, μπορώ να σας πω ότι αφενός έχει ωφεληθεί βεβαίως από την αριστεία η χώρα μου, ταυτόχρονα όμως ε, ανησυχούμε ε, για την πρόθεση της αριστείας. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν και η δική σας έκθεση και η έκθεση Λαμή μας δίνει πολύ καλές ιδέες για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μέσω της αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων ή και άλλων ταμείων. Αυτό που ε, θα ε, προσπαθήσουμε εμείς να επιτύχουμε είναι ε, σημαντικά και σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι έχουμε πολύ καλά έγγραφα πάνω στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε και από εκεί και πέρα μπορούμε να επικεντρωθούμε και στα θετικά αποτελέσματα που έχουν αποφέρει ε, οι διάφορες συμπράξεις ε, δημοσίου ιδιωτικού τομέα, τι επιτεύγματα έχουν ε, καταφέρει να επιτύχουν ίδια, τα διάφορα κράτη-μέλη και από εκεί και πέρα να παραδώσουμε όλη αυτή την εμπειρία που θα έχουμε συλλέξει και στην επόμενη Προεδρία, τη Βουλγαρία. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου και ελπίζω πως όλες οι παρατηρήσεις που κάναν οι συνάδελφοι και όλα τα ερωτήματα θα είναι σημαντικά για την Προεδρία σας και θα τα λάβετε δεόντως υπόψη τη στιγμή που θα οδηγείτε εσείς την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη θέση σας στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αρχική σας παρουσίαση, για το γεγονός πως μας τιμήσατε με την παρουσία σας στο Κοινοβούλιο και εμείς είμαστε πολύ ανοιχτοί στο μέγιστο της συνεργασίας, όπως προτείνατε και στην αρχή με τα όσα μας είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ και κάθε επιτυχία. Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να περάσουμε τώρα στο σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε τον κύριο Πέτρεσεν που είναι ο εισηγητής για το θέμα αυτό, που είναι ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ιθμιστικών Αρχών Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ε, μία αναδιατύπωση που έχει ο σκοπό να περιγράψει τις νέες αρμοδιότητες της ρυθμιστικής αυτής αρχής, όπως επίσης τα όσα γίνονται σε σχέση με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και πρέπει να σας πω ότι έχουμε 36 τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσης. Και κυρίως για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την αρχή αυτή. Οπότε, αυτό έχει να κάνει ο εισηγητή μας, σε γενικές γραμμές και τώρα μπορώ να σας ζητήσω αγαπητέ συνάδελφε, να μας παρουσιάσετε τα όσα έχετε να πείτε πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. King, uh, the shadows, uh, Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους Σκιώδης τα έχουμε συζητήσει. Είναι ένα τεχνικό και αρκετά περίπλοκο ζήτημα και οργανώσαμε ένα σεμινάριο για να μάθουμε περισσότερα για την πρόταση και τα συγκεκριμένα στοιχεία και πιστεύω ήταν πολύ ενδιαφέρον για όλο μας να ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι διάφορες πλευρές που εμπλέκονται στο θέμα. Χρειαζόμαστε μια εσωτερική αγορά για την ενέργεια και τα πλεονεκτήματα ήταν πολλά για τους καταναλωτές, για τις εταιρείε όπως επίσης και για τον ίδιο τον πλανήτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει πως αν έχουμε επαρκή παραγωγή ε, ενέργειας θα εξοικονομήσουμε 7,5 δις ευρώ κάθε χρόνο. Όμως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εσωτερική αγορά ενέργειας. Αντίθετα, δεν έχουμε καταφέρει ούτε τους πιο εύκολους καρπούς να συλλέξουμε, που είναι να προσφέρουμε κάποια πλεονεκτήματα φθηνή ηλεκτρική ενέργεια στου καταναλωτές, γιατί δεν έχουμε ελεύθερη ροή ηλεκτρικής ενέργειας διασυνοριακά. Είναι σπάνιο το φαινόμενο και δεν μπορούμε να στείλουμε φθηνή ηλεκτρική ενέργεια εκεί που είναι ακριβή. Πολύ συχνά ο βρόχος μεταξύ ε, Γερμανίας και Δανίας, το λέω, ε, είναι ε, μπλοκαρισμένος και χάνονται περίπου 13 εκατομμύρια το χρόνο και αν δείτε παντού στην Ευρώπη οι προκλήσεις είναι οι ίδιες και αυτό θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε και να πετύχουμε εξοικονόμηση μέσω μιας λογικής αναδιάταξης. Τώρα στην Επιτροπή μας πολύ συχνά λέμε πως θέλουμε η αγορά να λειτουργήσει. Αν όμως για να λειτουργήσει η αγορά χρειαζόμαστε ρύθμιση, τότε θα πρέπει η ΕΝΗΣΑ μαζί με τη ρυθμιστική αρχή που έχουν συντάξει κώδικες για τα δίκτυα και που έχουν προσπαθήσει να πετύχουν μεγαλύτερη τυποποίηση, να έχουν την ευκαιρία να λάβουν περισσότερες πληροφορίες που θα τους επιτρέψουν και θα μας επιτρέψουν να περάσουμε στην εφαρμογή, γιατί εκεί είναι το κλειδί της επιτυχίας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε να τονίζουμε το πόσο σημαντική είναι η επικουρικότητα και να εξασφαλίσουμε πως οι αποφάσεις λαμβάνονται στο σωστό επίπεδο. Και αυτό ακριβώς σημαίνει ότι περισσότεροι περιφερειακή συνεργασία. Γιατί αν δεν υπάρχει, τότε η εθνική TSO και τα κράτη-μέλη τι κάνουν, προστατεύουν τις δικές τους αγορές. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια ισχυρή περιφερειακή διάσταση μαζί με τα ROC, αυτά δηλαδή τα περιφερειακά κέντρα και εδώ στο σημείο αυτό πρέπει να επιμείνω. Εγώ μίλησα με TSO που μαζί είπαν με αυτά τα κέντρα θα ε, διακυβέσουν τις, ε, τη λειτουργία μας. Μα σας παρακαλώ συνάδελφοι, διαβάστε, σας παροτρύνω την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με πάρα πολλέ παρανοήσει. Είναι πάρα πολύ τεχνικό ο φάκελο και θα ήθελα να συζητήσουμε ανοιχτά, δίκαια, χωρί παρανοήσει, αυτό το πότοσο σημαντικό θέμα. Τώρα για τη ρυθμιστική αρχή να σας πω πως εγώ παρουσίασα διάφορα μέτρα στην έκθεσή μου και για τις αρμοδιότητες του Διευθυντή. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να τις ενισχύσουμε και να του επιτρέψουμε ή να τις επιτρέψουμε να ζητήσει από τι περιφερειακές ρυθμιστικές αρχές να παραπέμπουν στην αρχή προτάσει προ απόφαση. Και σε περίπτωση που υπάρχει απτό, τη συνέπεια στην εσωτερική αγορά συν, ηλεκτρικής ενέργειας. Ξέρουμε πως αυτή τη στιγμή αυτή η αρχή έχει περιορισμένους πόρους ε, και είναι πολύ λιγότερο από αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Άρα λοιπόν μία τέτοιου είδου υπηρεσία, μια τέτοιου είδου αρχή, για να είναι λειτουργική χρειάζεται σταθερή χρηματοδότηση, άρα λοιπόν θα μπορεί να συλλέγει και τέλη για κάποιε υπηρεσίε που προσφέρει. Είναι επίση σημαντικό το Διοικητικό Συμβούλιο τη αρχή να δρά προ το συμφέρον του κοινού και όχι κατόπιν πολιτική υπόδειξη. Και θα πρέπει να μην έχουμε υπερβολικά εξόδα... Ε, όταν προσπαθούμε να καταλήξουμε σε αποφάσεις επειδή ακριβώς οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ε, δεν θέλουν να μετακινηθούν σε κάποιο θέμα. Το έχω ζητήσει με του συμμαντέλου. Εκεί χρειάζεται προσπάθεια. Και επίση θα πρέπει να λογοδοτεί η αρχή αυτή προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι όπω προβλέπει ο τρέχον κανονισμό λειτουργία τη. Όλα αυτά πιστεύω πω θα την φέρουν την αρχή αυτή προ την σωστή κατεύθυνση και θα αποτελέσει και ένα καλό βήμα έτσι ώστε να πετύχουμε την πραγματική εσωτερική αγορά. Και εμείς ως πολιτικοί αυτό το οφείλουμε στον Ευρωπαίο πολίτη. Είναι ένας χώρος στον οποίο η Ευρώπη θα περιμένει από εμά να προσφέρουμε λύσεις που θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές και σε πλεονεκτήματα. Ας Κάνουμε τη δουλειά μας λοιπόν. Με χαρά θα ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων από τους υπόλοιπους σκιώδεις και με μεγάλη χαρά αναμένω να συνεχίσουμε την καλή δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα με συναδέλφους. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση, για την ομιλία σας, για να ανοίξουμε τη συζήτηση. Πόχε τώρα, ως ο από τους σοσιαλιστέ. Δεν υπάρχει ΕΛΚ. Κανένα πρόβλημα. Πολύ ωραία. Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί, ευχαριστώ τον Μόρτεν για την έκθεσή του και την αυτορία. συνεργασία. Η αναδιατύπωση έχει δύο πτυχές. Αυτά με τις αρμοδιότητες της ESA. Τις δίνουμε περισσότερες αρμοδιότητες για διασυνοριακά ζητήματα. Και το δεύτερο αφορά τη λειτουργία των επιμέρους οργάνων. Η άποψή μου είναι ότι χρειαζόμαστε έναν ισχυρό οργανισμό με περισσότερες αρμοδιότητες, περισσότερες εξουσίες, δυνατότητες επιβολής, και το οποίο θα σημαίνει φτηνότερη ενέργεια για τους πολίτες. Ε, το ξαναλέω δεν είναι μόνο περί αρμοδιορίτων και εξουσιών, είναι και θέμα πόρων. Έχει σημασία ο οργανισμός να έχει στη διάθεσή του πόρους, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την εσωτερική αγορά. Χρειάζεται όμως και δυνατότητα λήψη αποφάσεων για να καλύπτει κενά στην νομοθεσία, για παράδειγμα. Πρέπει επίση να έχει τη δυνατότητα να εκδίδει δεσμευτικές και εφαρμόσιμες αποφάσεις για δραστηριότητε σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι ο οργανισμός επίσης πρέπει να έχει την δυνατότητα να υποχρεώνει διάφορους φορεί να συμμορφώνονται μέσω προστήμων που θα επιβάλλουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Ο οργανισμός επίσης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει πρόστιμα και απευθεία στην περίπτωση μη συμμόρφωσης. Έτσι λοιπόν. Ο οργανισμός αυτός εργασίας θα διαδραματίσει πραγματικό ρόλο στην αγορά. Πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες επίσης ψηφορία για την ανάδειξη του Συμβουλίου και πρέπει η Επιτροπή να άρει την υποχρέωση των μελών του Συμβουλίου να μην υπακούν σε πολιτικέ οδηγίες. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι πρώτον ε, ε, έλλειψη πόρων, ο ACER, ο εργασία των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, πρέπει να έχει περισσότερε δυνατότητε. Δεύτερον, όσον αφορά την ψηφορία, την ανάδειξη του Συμβουλίου. Αυτό πρέπει να γίνεται με απλή ψηφορία παρά με πλειοψηφία δύο τρίτων. Δεδομένου ότι κάθε κράτος έχει μία και μόνη ψήφο. Τώρα το αν το Συμβούλιο θα επακούσει πολιτικά και αυτό είναι μια ε, άλλη ιστορία, αλλά αυτό είναι που θα καθαρίσει την απόδοση και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Χρειάζεται πλέον διαφάνεια, χρειάζεται λογοδοσία τόσο σε επίπεδο Acer όσο και σε επίπεδο μελών από τις χώρες μέλη. Πρόεδρος επόμενος ομιλητής είναι ο δικαστάς του κ. Χένκελ, ο σκιώδης της ECR. Παρακαλώ. Πρόεδρε, Ευχαριστώ. Ο σκιώδης μας δυστυχώς δεν μπορούσε να έρθει σήμερα, οπότε θα παρουσιάσω τη θέση του. Ευχαριστούμε λοιπόν τον εισηγητή για την έκθεσή του. Πολύ θετική η ματιά του εναντί της προτάσεω της Κομισιόν. Έχουμε υποβάλει τροπολογίες. Η 5 μας βρίσκει σύμφωνος, γιατί σύμφωνα με την 5 θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε δεσμευτικούς κανόνες και να πετύχουμε συμμόρφωση με τον κώδικα. Οι δεσμευτικές αποφάσεις πρέπει να υλοποιούνται από τις εθνικές αρχές και το πενετήματος του Acer που θα μπορεί επίση να ζητάει στοιχεία και πληροφορίε από τι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ εντό των πλαισίων τη εντολή του και βεβαίω ε, στα πλαίσια διαφάνειας και κυριότητας της χοντρικής αγοράς. Δεν θέλουμε συγκεντρωμένες, υπερσυγκεντρωμένες αγορές, ούτε έλεγχο, θέλουμε μια απελευθερωμένη αγορά, ώστε να διατίθεται την Ευρώπη ρεύμα σε χαμηλές τιμές. Υπάρχει και μια διασυνοριακή πτυχή. Εδώ για άλλη μια φορά χρειαζόμαστε Περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη εποπτεία από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό για την επίτευξη ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας του φωτισμού, για να μην μιλήσουμε και για τις τιμές. Αυτά δεν μπορεί να κάνει η σημερινή Acer, ο σημερινός Acer. Γι' αυτό και θα προτείνουμε έναν αυξημένο προπολισμό. Συγγνώμη για την μακροσκελή παρουσίαση, αλλά αυτά ήθελα πει ο και μετέφερα εγώ. Και στο μας. Ευχαριστώ, Ο Ταβόρ δεν μπόρεσε να έρθει, οπότε θα σας δώσω εγώ μια σύνοψη της θέσης μας. Ως πράσινοι θεωρούμε ότι δεν υπάρχει άλλος οργανισμός με τόσο μεγάλη ε, θετική ε, ε, αναλογία επενδύσεων και αποτελέσματος. Με κάποια πραγματικά λίγα εκατομμύρια μπορείς να δρέψεις καρπούς εκατοντάδων εκατομμυρίων. Αυτό βέβαια είναι και το πρόβλημα κατά μία έννοια. Γιατί στον Acer ε, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό είναι πολύ σημαντικό να ε, αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Εγώ ε, συμφωνώ να διατηρηθεί το όνομα ROC, γιατί χρειάζεται μερικές φορές να ασκήσεις κάποιους κραδασμούς ενδεχομένως για να διατηρηθεί μια ορμή. Αυτό που ε, όμως για να είμαστε ε, ειλικρινείς είναι ότι υπάρχει μεγάλη αντίθεση μεταξύ του Acer και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και αυτό ε, πολλές φορές ε, το επέτεινε το πρόβλημα αυτό η έλλειψη διαφάνειας. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να δοθούν περισσότερε αρμοδιότητες στον Acer, αλλά πρέπει να δούμε αν οι εσωτερικοί κανόνες διαφάνειας πραγματικά ε, αντιστοιχούν ε, στην σημασία αυτού του ευρωπαϊκού οργανισμού. Δεύτερον, νομίζω ότι ε, ο Acer έχει ενοχλήσει διάφορους εμπλεκόμενους φορείς το να γίνεται μια ε, αναδρομική ακύρωση ε, αυτής της, της ε, κατά προαιρεότητα εισαγωγής της ενέργειας από ΑΠΕ με εξέπληξε. Πραγματικά μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι οι ρυθμιστικές αρχές ε, έχουν χάσει το στόχο. Δεν κάνουμε εμπόριο για το εμπόριο απλά και μόνο σε αυτό σκοπό, αλλά γιατί μέσω της αγοράς και του εμπορίου μπορούμε να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Στόχος πρέπει ε, η ΑΠΕ να, πρέπει να είναι η ΑΠΕ να φτάσουν στο 100%. Και τέλος που αποτελεί και ερώτημα προς την Κομισιόν. Υπάρχει κάτι παράδοξο. Πρόκειται για τις ε, εκλογικές διαδικασίες. Έχουμε ένα λόμπι το οποίο ε, ε, έχει το όνομα ΣΥΑ και από εκεί και πέρα βλέπουμε να υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ ενός λόμπι και του, του Διοικητικού Συμβουλίου των Ρυθμιστικών Αρχών. Το CER για μένα είναι ένα λόμπι των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και κατά τη γνώμη μου δεν είναι σωστό να ε, υπάρχουν άτομα και να ακολουθούνται εκλογικές διαδικασίες όπου ε, μόνο, ε, μπορεί να υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος. Γιατί αυτό δημιουργεί μια σύγχυση μεταξύ του χαρακτήρα του ενός επίσημου ευρωπαϊκού οργανισμού και του χαρακτήρα ενός λόμπι. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι το CER θα πρέπει να έχει πρόεδρο και από εκεί και πέρα ε, ο Οργανισμός των Αθηνιστικών Αρχών ε, θα έχει έναν άλλο πρόεδρο. Διότι αλλιώς θολώνουν τα όρια ε, μεταξύ αυτών των δύο διακριτών κατά τη γνώμη μου φορέων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σιλικιώτης εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Πρόεδρε, ε, αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μόρτε για την συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα. Ε, για την ομάδα μας στην Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά είναι ξεκάθαρο Καθώ ο ΕΣΕΡ δεν είναι ευρωπαϊκός οργανισμός, δεν είναι agency αλλά μια πλατφόρμα συνεργασίας των εθνικών ρυθμιστικών αρχών εξορισμού δεν μπορεί και δεν πρέπει να διαμορφώνει στρατηγική. Έπειτα, μέχρι σήμερα η Ένωση απέτυχε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ενορχιακού εφοδιασμού που έχουμε στην Ένωση και να άρει την ενεργειακή απομόνωση στην οποία βρίσκονται κράτη και περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ιδιαιτερότητε λοιπόν των κρατών μελών, τα ιδιαίτερα προβλήματα και ανάγκε που έχουν, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη. Εν τούτης, δυστυχώς, οι προτάσεις που αναπτύσσονται ε, στην πρόταση της Κομισιόν και υποστηρίζονται και από τον συνάδελφο συγητή Πέτερσεν οι αυξημένε αρμοδιότητε των Acer καταστρατηγούν τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών στη διαμόρφωση τη ενεργειακή του πολιτική και υπομονεύουν το σημαντικό ρόλο που παίξαν μέχρι σήμερα και παίζουν οι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ. Ιδιαίτερα προβληματική για μα είναι η πρόταση του άρθρου 43, πω το Διοικητικό Συμβούλιο του Acer θα εγκρίνει στρατηγική για τις σχέσεις με τρίτες χώρες. Ο ΕΣΕΡ δεν είναι πολιτικό όργανο και δεν πρέπει να λάβει τέτοιες υπερεξουσίες. Η όρη συνεργασία με τρίτες χώρες είναι απόφαση των κρατών μελών και αφορά μονάχα εκείνες τις τρίτες χώρες που έχουν υιοθετήσει και εφαρμόζουν τον κεκτημένο της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος κατόπιν ένα συμφωνιών με την Ένωση. Δεν μπορεί λοιπόν ο Acer να αποφασίζει αυθαίρετα βάσει άλλων κριτηρίων για τόσο σημαντικά θέματα. Κλείνοντα, θέλω να αναφερθώ στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο που είναι και το κύριο όργανο λήψη αποφάσεων του Acer. Η αντικειμενική λειτουργία του και η αντιπροσωπευτική συμμετοχή όλων των μελών του είναι ζωτική σημασία. Για, τον λόγο, για τον λόγο αυτόν εμεί την τροποποίηση που προτείνεται στο άρθρο 23 όσον αφορά του κανόνε τη εφορία, ε, πριν χρειαζόταν τα δύο τρίτα για να περάσει μια απόφαση τότε απαιτείται απλή πλουσφία, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και υπονομεύει την λεπτή ισορροπία της αντιπροσωπευτικής συμμετοχής και θεωρώ, ενώ δεν φαίνεται τούτο, ότι τελικά αυτό που θα είναι σε βάρος κυρίω των μικρών κρατών μελών της Ένωσης ε, γιατί ξέρουμε πώς λειτουργούν ε, τα ζητήματα των συνεργασιών ε, και ε, σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις. Ε, και είναι στη βάση αυτών των παρατηρήσεων που θα καταθέσει η τροπολογίες η δική μου πολιτική ομάδα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you very Ευχαριστώ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Διευθυντά Μπόρχαντ. Όπως πάντοτε άλλωστε όταν συζητούμε τα ζητήματα του πακέτου ενέργειας. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που σας έχω κουράσει με την παρουσία μου. Όχι, όχι, λέει ο Πρόεδρος. Αντίθετα, εμείς ε, χαιρετίζουμε τη συνεργασία και είναι απολύτως απαραίτητη μαζί σας. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να χαιρετήσω την ε, έκθεση του κυρίου Πέτρισεν και της τροπολογίες. Όχι μόνο γιατί υποστηρίζει την πρόταση Κομισιόν, κάτι για το οποίο βεβαίως είμαστε ευγνώμονες, αλλά και διότι στις τροπολογίες με, κατά κάποιο τρόπο ενισχύει την δική μας πρόταση. Σε ένα σημείο πρέπει να σας πω ωστόσο ότι είστε λιγότερο φιλόδοξο από εμάς. Και θέλω να επικεντρωθώ σε ακριβώς αυτό το σημείο. Να αναφερθώ βεβαίως και σε ζητήματα που θεωρώ ότι ε, ενισχύεται τη δική μας θέση. Είστε λιγότερο φιλόδοξοι όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ε, βλέπετε την συμμετοχή του Acer στην ε, λήψη αποφάσεων για τις μεθοδολογίες που ακολουθούνται σε περιφερειακό επίπεδο. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που προέρχονται από τους κώδικες δίκτυων. Πρώτον, δίνεται, ε, δυνατότητα στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και αφού αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, τότε δίνεται δυνατότητα αυτή στον Acer. Επειδή λοιπόν δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική αυτή η διαδικασία, θεωρήσαμε ότι είναι πολύ καλύτερο να, δοθ, να λαμβάνονται αυτές οι περιφερειακές αποφάσεις από τον Acer σε ε, σχετική υποεπιτροπή που θα αποτελείται από εκπροσώπους των ε, ε, εκάστοτε περιοχών. Αυτό όμως είναι και το μόνο σημείο στο οποίο βλέπω ότι υπάρχει ένα χαμηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας από εμάς. Αντίθετα, τα σημεία όπου στην πραγματικότητα με τις προτάσεις σας ενισχύεται την πρόταση κομμισιών και εσείς και οι συνάδελφοί σας είναι ότι πρώτον ε, δεν βρίσκεται ε, τίποτα στη δική μας πρόταση σχετικά με τη χρηματοδότηση. Άκουσα πολύ υποστήριξη εδώ ότι ε, στο, στη δυνατότητα του Acer να επιβάλλει τέλη. Αυτό πράγματι είναι ένας τρόπος για να ενισχυθεί οικονομικά η κατάσταση του Acer. Πρέπει ωστόσο να δούμε πολύ προσεκτικά τη διατύπωση που θα χρησιμοποιήσουμε, διότι αυτή η διατύπωση θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται πλήρω με του ε, δημοσιονομικού κανόνε, καθώ και με το νομικό πλαίσιο εντό του οποίου οι οργανισμοί γενικά καλούνται να δραστηριοποιηθούν. Παρ' όλα αυτά, είμαι βέβαιο ότι μπορούμε να βρούμε αυτή τη διατύπωση ώστε να δίνεται δυνατότητα ε, τελών ε, εντός του νομικού και δημοσιονομικού ε, πλαισίου που ισχύει. Αν χρειαστεί βεβαίως ε, μπορούμε και να σας συνδράμουμε σε αυτό. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι παραβλέψαμε εμείς αλλά όχι εσείς και σας συγχαίρω γι' αυτό είναι το γεγονός ότι δίνεται νέες αρμοδιότητες στον Acer προκειμένου να απαιτεί εκείνος ε, τις απαραίτητες από, τα, από τους, ε, από τους ε, ε, TSO, οι οποίοι πολλές φορές στο παρελθόν δεν ήταν ιδιαίτερα πρόθυμοι να δίνουν σχετικές προφορίες. Το μόνο μου αίτημα είναι να επεκταθεί αυτή η, το μόνο μου αίτημα είναι να μην επεκταθεί αυτό στο, στους ένσω του φυσικού αερίου διότι σε αυτή την περίπτωση ε, στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε μια διαδικασία ε, αντικατοπτρισμού δηλαδή του, της ροής του φυσικού αερίου. Εδώ νομίζω ότι κάπως αρχίζετε και τα μπλέκετε. Δεν σας ασκώ κριτική, απλά το επισημενο ως ε, ένα υπαρκτό θέμα που εντόπισα στην έκθεσή σας. Επίσης, ενισχύεται και τον ε, ρόλο του Acer όσον αφορά την συμμόρφωση. ζητήσατε οι Εθνικέ ρυθμιστικέ αρχές να συμμορφώνονται με τι αποφάσει του Acer. Με αυτό δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τροπολογία 4. Στην τροπολογία 5 όμως πηγαίνατε λίγο παραπέρα. Θεσπίζοντας δεσμευτικές αποφάσεις του Acer προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις νομικές πράξει. Εδώ η μόνη μου επιφύλαξη είναι η εξή. Αυτό δεν είναι ε, αποκλειστική αρμοδιότητα της Κομισιόν ως θεματοφύλακα ε, της ε, ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Μήπως δεν πρέπει να απονεμηθεί, να αποδοθεί ένα τέτοιος ρόλος σε οργανισμό, το να εξασφαλίζεται δηλαδή η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Νομίζω ότι είναι κάπως οριακό αυτό που προτείνεται εδώ από αυτή την άποψη. Επίσης, ενισχυμένη κανονιστική εποπτεία, αυτό που είπε ο κύριος Τούρμες Ρόξ, από το, σήμερα το πρωί όμως πλέον εγώ αποκαλώ, ε, ε τους αποκαλώ RCC. Ε, υπάρχουν βεβαίως και τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα που συζητήσαμε σήμερα το πρωί. Είναι το λογικό επόμενο βήμα. Όταν υπάρχουν συνέργειες σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη παρακολούθηση και εποπτεία. Υπάρχουν πάρα πολλοί ανησυχίες οι οποίες έχουν εκφραστεί, οι οποίες μάλιστα θα διασκεδαστούν αν συσταθούν αυτά τα ρυθμιστικά συντονιστικά ε, κέντρα, ακριβώς γιατί θα έχει εξασφαλιστεί και η υποπτία τους. Τα υπόλοιπα σας τα είπα σήμερα το πρωί, ως προς την αναγκαιότητα να, υπάρχει να υπάρχουν αυτή, αυτά τα όργανα για την περιφερική συνεργασία. Τέλος, να απαντήσω στο ερώτημα του κυρίου Τούρμες προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των Προέδρων ε, του Διοικητικού Συμβουλίου των Ρυθμιστικών Αρχών και όπως είπατε σωστά, ταυτόχρονα του, ε, του Προέδρου του ΣΥΑ, ΣΥΑ, που είναι ιδιωτικός οργανισμός. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας ε, στο ΣΥΑΡ και έχουμε πει ότι η Κομισιόν δεν θα αποδεχθεί την προβλεπόμενη εκλογική διαδικασία όπου στην πρώτη φάση η ΣΥΑΡ ορίζει τον πρόεδρό της και στη συνέχεια το ίδιο πρόσωπο ε, αναλαμβάνει τη θέση του, του, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό ε, και απλά έρχεται και επισφραγίζεται μια προηλημένη απόφαση. Αν πράγματι συμβαίνει αυτό θα καταγγείλουμε την ε, εκλογή αυτή. Δεν πρόκειται να τα αποδεχτούμε. Πράγματι συμφωνώ μαζί σας κύριε Τούρμες ότι το καλύτερο θα ήταν να είναι δύο ξεχωριστά διαφορετικά πρόσωπα. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε. Αυτό που μπορούμε όμως να επιβάλλουμε είναι ότι η εκλογή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να προηγείται και μάλιστα να γίνεται με ε, πλειάδα υποψηφίων. Στη συνέχεια, άμα θέλουν στον ιδιωτικό του οργανισμό να ε, εκλέξουν το ίδιο πρόσωπο, ας το κάνουν. Όμως η σειρά πρέπει να είναι η σωστή. Πρώτον ε, Board of Regulators και στη συνέχεια ε, ο κάθε ιδιωτικός οργανισμός μπορεί να επιλέγει ε, τον, τον πρόεδρό του αυτόνομα. Αν υπάρχει οποιαδήποτε απόκληση, παρέκκληση από αυτή τη διαδικασία που περιέγραψα, εμείς θα την καταγγείλουμε και θα προσφύγουμε κατά της. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε και τη δική σας θέση και θα ήθελα τώρα να ζητήσω για τις τελευταίες παρατηρήσεις του συνάδελφου κύριο Πέτερσταν. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους συναδέλφους για κάθε μία από τις παρατηρήσεις που έκαναν. Και να σας πω πως αισθάνομαι πολύ αισιόδοξο για τη δυνατότητα που έχουμε να πετύχουμε μια ευρία πλειοψηφία, γιατί αυτός είναι βέβαια και ο στόχος μας. Πιστεύω δηλαδή πως είναι πολύ σημαντικό σε όλους τους φακέλους που αντιμετωπίζουμε στο πακέτο αυτό είναι να έχουμε ευρία πλειοψηφία όπως κάνουμε γενικά στο Κοινοβούλιο για να μπορούμε μετά να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο και να είμαστε στο δυνατόν πιο ισχυροί. Ε, συνάδελφε Πόχε, σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια. Νομίζω πως υπάρχει κοινό τόπος στον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Τοσινόφσκι ε, και την ECR ε, για την στήριξη που μας προσφέρουν και να σας πω πως ε, έχω αισιοδοξία τώρα. Θα τα καταφέρουμε. Και κύριε Τούρμες τώρα, δεν νομίζω πώς θα μπορέσω να συμφωνήσω με το όσο προτείνει ο κύριος Σίλη και ότι θα τον προσπαθήσω. Θα δω τι μπορούμε να κάνουμε στις διαπραγματεύσεις και τέλος για τις παρατηρήσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σας πω πως βέβαια με εκνευρίζει όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει πως δεν είμαστε εμείς τόσο φιλόδοξοι ως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να δούμε μήπως το διορθώσουμε αυτό στις διαπραγματεύσεις και για τις νομικές λεπτομέρειες σίγουρα πρέπει να συμμορφωθούμε με τη νομική βάση για να εξασφαλίσουμε πως αυτά θα γίνουν σωστά. Και χαίρομαι που μου κάνετε κάποια πρόταση να μας βοηθήσετε να βρούμε κάτι το οποίο είναι εύχριστο και σίγουρα θα έχουμε μια καλή νομική βάση. Ξέρετε και εσείς που το χρονοδιάγραμμα λέει προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών μέσα Σεπτεμβρίου. Οπότε, στις διακοπές σας, εσείς συνάδελφοι, ελπίζω να εμπνευστείτε εκεί που αναπάβεστε και να γυρίσετε γεροί και δυνατοί με στο Σεπτέμβριο με τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ, όπως σας είπα είμαι αισιόδοξο. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο τέλος θα δούμε πόσο φιλόδοξο ήταν το Συμβούλιο. Τώρα ακόμα δεν το ξέρουμε. Και δεν ξέρουμε πόσο μακρά, μακριά στοχεύει. Τώρα μπορούμε να πούμε πως Προθεσμία τελική 14 Σεπτεμβρίου για την υπολογή, υποβολή τροπολογιών. 14 Σεπτεμβρίου του 17, 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή, ευχαριστώ πολύ τους κοιόδης, ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους που πήραν μέρος στη συζήτηση και βεβαίως ευχαριστώ και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλη την ομάδα και βέβαια το Διευθυντή πρώτον από όλους. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, στο σημείο αυτό προχωρούμε στη συγκρότηση κοινή επιχείρηση βιομηχανικών βιοπροϊόντων. Ένας ΔΙΤ στα πλαίσια του άρθρου 187 είναι φάκελος διαβούλευσης και ο στόχος είναι αυτή η επιχείρηση όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να τους φέρει κοντά έτσι ώστε να συρισφέρουν στην προώθηση της Ευρώπης ως μεγάλος ανταγωνιστής για τα βιοπροϊόντα και τα βιοκαύσιμα στην αγορά. Σας το διάβασα έτσι γιατί έτσι μου το έχουν γράψει. Και έτσι γράφεται και στον κανονισμό. Η συγητής, το 14 ήταν ο κύριος Βαν Ρόι. Και βέβαια αυτή η κοινή επιχείρηση θα αρχίσει να, με συγχωρείτε, θα λειτουργεί για τέσσερα χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2024. Σήμερα έχουμε έναν εισηγητή που είναι ο κύριος Μυροσλάβ Πόχια. Συνάδελφε, σας ζητώ να μας κάνετε μία πρώτη παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα κι εγώ να σας ευχαριστήσω και να σας πω πως ήταν πολύ ευχάριστο και το απόγευμα, ήταν ωραία και εισαγωγή που κάνατε και αυτή η κοινή επιχείρηση θα αποτελέσει μία από επτά κοινές επιχειρήσεις που ξεκίνησε να λειτουργεί το 2015 τον Νοέμβριο και ο κανονισμός λέει θα λειτουργήσει για 10 χρόνια μέχρι το 2024. Στόχος να ενισχύσει τα βιοπροϊόντα και στην, στο χώρο της έρευνας και να εισάγει τις βιοτεχνολογίες και τα βιοκαύσιμα στην αγορά. Η έκθεση αυτή έχει να κάνει με τον τροποποιημένο κανονισμό έτσι ώστε να αλλάξει ο εσωτερικός μηχανισμός χρηματοδότησης. Συνολικός προϋπολογισμός 3,7 δις και τα χρήματα προέρχονται από τον ιδιωτικό κλάδο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ιδιωτικό κλάδος έχει φτιάξει ένα όχημα, έναν όμιλο που συνεισφέρει 0,7 δις ευρώ από τα 3,7. Και οι συνεισφορές αυτές είναι σε είδος κυρίως. Αλλά έχουμε και ένα 1,82 εκατομμύρια ευρώ για ε, τρέχοντα ε, λειτουργικά έξοδα και αυτές είναι οι συνεισφορές που γίνονται μέσα στο πρόγραμμα. Όμως, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα. Γιατί? Γιατί κάποιες εταιρείες συνεισφέρουν οικονομικά χωρίς να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε project. Δηλαδή, έχουμε την εταιρεία Α που βάζει μετρητά στην επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά για ένα σχέδιο το οποίο δεν έχει αναλάβει η επιχείρηση Α, αλλά η επιχείρηση Β. Και η επιχείρηση Β μπορεί να αποτελεί άμεσο ανταγωνιστή τη επιχείρηση Α. Οπότε καταλαβαίνετε πω οι επιχειρήσει δεν έχουν και ιδιαίτερη όρεξη να χρηματοδοτούν project τα οποία ενδεχομένω μπορεί ε, να ε, θέσουν ένα αμφιβόλο και την επιτυχία του προγράμματο και τι ίδιε επιχειρήσει και ιδιαίτερα να έχουν αρνητικέ επιπτώσει ανταγωνιστικά για τον κλάδο. Και αυτό φαίνεται από την τάση που έχουμε με τα νούμερα. Από τα 182 εκατομμύρια ευρώ, λιγότερο από 1 εκατομμύρια ευρώ ε, μπήκε σε αυτή την επιχείρηση με τον τρόπο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αλλάζει τον κανονισμό, κάνει μια τεχνική προσαρμογή που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να συνεισφέρουν ε, ανά project, δηλαδή είναι μια άμεση πληρωμή σε άλλους συμμετέχοντες του ίδιου ε, ομίλου ε, στο ίδιο project. Και αυτό προτάθηκε μετά από διαβουλεύσεις με τα μέλη αυτών των ομίλων, όπως επίσης και με την επιστημονική κοινότητα και με, τα με τους εμπλεκόμενους φορείς. Όλοι αυτοί ε, συζήτησαν το θέμα και κατέληξαν σε αυτή την απόφαση. Έχω κάνει μια απογραφή των προτινόμενων αλλαγών και θέλω να δω αν αυτέ οι αλλαγέ στη χρηματοδότηση θα δημιουργήσουν επιπλοκέ στο μέλλον ή όχι. Και στη βιομηχανία και αλλού. Και βασιζόμενο σε αυτή την αξιολόγηση που έκανα, τελικά θα στηρίξω την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό όλε αυτέ οι συμφωνίε και όλα τα προγράμματα να εφαρμοστούν με διάφανο τρόπο, με ανοιχτό τρόπο και έχω μάλιστα να κάνω και μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θέλετε εσεί, Αυτά τα 70 εκατομμύρια ευρώ που αυτή τη στιγμή ε, είναι ε, ε, στο απόθεμα τι θα τα κάνετε, θα προχωρήσετε σε διαγωνισμούς, θα στήσετε κάποια καινούργια project βιοτεχνολογικά, θα τα κρατήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις έρευνες που κάνετε συνάδελφοι και σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις προσπάθειες για να ε, μας δώσετε όλες αυτές τις πληροφορίες και να μοιραστείτε μαζί μας όλα τα στοιχεία τούτα. Νομίζω ότι θα πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς γνωρίζοντα όλα αυτά τα καινούργια που μας είπατε για αυτές τις κοινέ επιχειρήσεις που αποτελούν επαναλαμβάνω ΣΔΙΤ. Σας ευχαριστώ και πάλι. Εκ μέρους του ΕΛΚ έχουμε τον κύριο Γκάμπους. Έχετε το λόγο συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να πω στον κύριο Πόχελ πως η δουλειά που έκανε ήταν καταπληκτική και είμαι σίγουρος πως θα καταλήξουμε σε μια πολύ ικανοποιητική συμφωνία με τις τροπολογίες οι οποίες θα κατατεθούν. Πιστεύω πως τα είπε πολύ καλά και μας εξήγησε με μεγάλη σαφήνεια ποιο είναι το πρόβλημα, το ουσιαστικό πρόβλημα και ποιες είναι οι δυσκολίες αυτή τη κοινή επιχείρηση για τη βιομηχανία βιοπροϊόντων και ποιε είναι οι δυσκολίε που αντιμετωπίστηκαν μέχρι σήμερα. Δεδομένου ότι έχουμε πολλά συμφέροντα και γενικότερα συμφέρον Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσουμε αυτά τα προϊόντα βιοτεχνολογίας και για να καταθέτουν οι βιομηχανίε βιομηχανίες τις του όπως έχει προταθεί, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιήσουμε το αρχικό κείμενο και να δώσουμε τη δυνατότητα οι χρηματικές εισφορές να γίνονται σε επίπεδο project. Γιατί τώρα αυτό που γίνεται είναι σε επίπεδο προγράμματος. Αυτή είναι μια λύση που νομίζω ότι θα λύσει το πρόβλημα και θα πετύχουμε τους στόχους μας, τους αρχικούς μας στόχους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει πως με την τροποποίηση αυτή θα αποφύγουμε κάποιες βλαβερές συνέπειες σε συνεργασίες που έχουμε ε, σε όλη την αλυσίδα συνεργασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, δύο προϊόντων, τα αποτελέσματα της έρευνας των ε, ερευνητικών κέντρων κτλ. Και αυτή είναι η βασική μας, η βασική μας υποχρέωση, ακριβώς να προωθήσουμε το ρόλο της μικρομεσαίας επιχειρήσης στον χώρο της βιοτεχνολογίας, έτσι ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τεχνολογικά αλλά και οικονομικά να προοδεύσει. Αλλά θέλω να δώσω μια μικρή χρειά, γιατί βέβαια όλα θετικά αυτά προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά μία ε, προσαρμογή του κανονισμού, μία τροποποίηση θα πρέπει να συνοδεύεται με δημόσια διαβούλευση ανοιχτή, διάφανη όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Έτσι ώστε να γνωρίζουν καλύτερα και οι Ευρωπαίοι πολίτε. Δηλαδή, χρειαζόμαστε να δούμε μία επιπτωσιακή μελέτη λεπτομερή και καταλαβαίνουμε ότι δεδομένη τη χρονική πίεση για να γίνει αυτή η τροποποίηση του κανονισμού δεν ακολουθήθηκαν όλε οι διαδικασίε τι οποίε μόλι προανέφερα. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να ζητήσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επόμενη φορά που θα κάνει κάτι τέτοιο να συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσει που έχουμε δημιουργήσει έτσι ώστε οι διαδικασίες να είναι ανοιχτέ και διάφανες στο μέτρο του δυνατού. Και θα κλείσω λέγοντας, ευχαριστώντας τον εισηγητή για όλη τη δουλειά που έκανε. Σας ευχαριστώ κύριε Πόχ και είμαι σίγουρος πως με τις τροπολογίες που θα καταθέσουμε η δουλειά που θα κάνουμε θα είναι εξαιρετική και θα καταλήξουμε σε μια πολύ θετική συμφωνία. Mr. Fox, Ευχαριστώ. Ο κ. Φόξ, που σαν τον κ. Πρόεδρε, η κυρία δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ. Ζητώ συγγνώμη από τους βουλευτές, πρέπει να φύγω για την έκονα αμέσως μόλις τελειώσει την ομιλία μου. Εμείς ε, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας ε, γιατί αυτή η προσπάθεια θα μειώσει τα έξοδα Ήδη παρόμοιες κοινοπραξίες λειτουργούν ικανοποιητικά και σύμφωνα με την ανάλυση της Κομισιόν ε, φαίνεται ότι η PBI θα μπορέσει και αυτή με αυτές τις συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις να πάει πολύ καλά. Πρέπει να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του ιδιωτικού τομέα και να βελτιώσουμε την δουλειά του BIC και του BBI. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία συνεργασία και ιδιωτικού τομέα. Αυτό θα αποφέρει βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων που έχουμε στη διάθεσή μα και θα ε, βελτιώσει γενικότερα τον τομέα. Κυρία Φανπόσερ, θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την έκθεσή του και η ομάδα μα η ECR προσβλέπει σε περαιτέρω συνεργασία. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συναδελφέ. Φυσικά, μιλήσατε εκ μέρου τη ECR. Ε, και τώρα να ακούσουμε την Αλντέρα, να ακούσουμε τους Κυρία Μάισνερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή και μπορώ να σας πω ότι συμφωνώ με τα όσα είπε ο συνάδελφος από το ECR. Γενικά θεωρώ ότι ε, είναι πραγματικά πολύ αξιολογή αυτή η πρωτοβουλία κάτι που βγαίνει, προκύπτει και από τις ε, γνωμοδοτήσεις Κοντ και Μπάντζ. Εμείς βεβαίως καλούμαστε να κάνουμε το πιο λεπτομερές έργο. Πάντως ε, το να προσθεθεί ε, μία ακόμα μέθοδος είναι κάτι πολύ θετικό στις ήδη υπάρχουσες, ακριβώς γιατί πρόκειται για έναν κλάδο ταχαίως αναπτυσσόμενο και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διευκολυνθεί η ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξή του. Στην πραγματικότητα δηλαδή ε, απλοποιούμε διάφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες και αυτό πάντοτε είναι θετικό. Όπως είπε και ο κύριος Φόξ, ε, αυτό ήδη διαπιστώθηκε ότι είχε θετικά αποτελέσματα και στον τομέα των ε, καινοτόμων φαρμάκων. Άρα έχει ε, διαπιστωθεί στην πράξη ότι πρόκειται για μια θετική διαδικασία. Γενικά είναι σημαντικό το γεγονός ότι συμφωνούμε ότι ο κλάδος αυτός θα έχει πολύ μεγάλη σημασία στο μέλλον. Μιλούμε και για ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ε, χρήση νέων υλικών και της, ε, της βενζίνης. Αυτό ε, είναι ένα στοιχείο ε, που διευκολύνει, συμβάλλει στην γενικότερη ανάπτυξη των ΑΠΕ. Φυσικά αυτό σημαίνει ότι ε, δεν έχουμε καθόλου αμφιβολίες, καθόλου ερωτηματικά. Αντίθετα προσβλέπουμε στην ε, ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ μας και με τον εισηγητή προκειμένου να ενισχύσουμε και να ε, προωθήσουμε την πρόταση αυτή της Κομισιόν. Ε... Ευχαριστώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Διευθυντής Μοναδάς κ. από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνα, Τεχνολογία και Ανάπτυξη. Το πλήρες όνομα της Γενικής Διεύθυνσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την εξαιρετική του ανάλυση. Δεν έχω νομίζω να προσθέσω πολλά. Ίσως μόνο να τονίσω την σημασία του τομέα που υπογράμμισαν διάφοροι προλαλήσαντες. Η βιομηχανία των βιοπροϊόντων αναπτύσσει τεχνολογίες που αποτελούν καταλήτη για πολλές, ή πολλές τομείς τις ανεώσιμες, ε, τα πλαστικά, τη χημική βιομηχανία, την προσπάθεια να παραγάγουμε προϊόντα ουδέτερα σε άνθρακα, ε, απόβλητα και πολλά άλλα προϊόντα. Και σε πολλούς άλλους τομείς, επαναλαμβάνω, ε, τρόφιμα, για μια κυκλική οικονομία, για περισσότερη ανακύκλωση. Είναι τεράστια σημασία του τομέα. Τα λοιπάσματα και ούτω καθεξής. Αυτά για να ξεκαθαρίσω πόσο, μεγάλο, πόσο μεγάλη σημασία έχει τομέα. Κάποιος ρώτησε ε, τον κύριο Πόχ, τι θα κάνουμε με τα 70 εκατομμύρια που περιμένουν αυτή τη στιγμή. Η Κομισιόν σε όλη την αφορά προστάτευσε τώρα τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα πρώτα χρόνια διαπιστώνουμε ότι δεν είχαμε χρηματοδοτήσει σε επίπεδο προγράμματος, όπω το είπε ο κ. Η βιομηχανία δεν θέλει να χρηματοδοτεί τον ανταγωνισμό. Οπότε μετακυλήσαμε τον προπολογισμό σε κατοπινές χρονιές και στη συνέχεια συνειδητοποίησαμε επίση ότι η βιομηχανία είχε θέματα. Ε, γι' αυτό και υποβάλαμε τροπολογίες Ελπίζω ότι το προηγείο φέτος αυτή θα υλοποιηθεί, θα εφαρμοστεί στην πράξη. Θα αξιοποιήσουμε το εργαλείο των διαγωνισμών και ότι τα πράγματα από εδώ και πέρα θα προχωρήσουν όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Έτσι, τα 77 εκατομμύρια θα επέλθουν στον προορισμό του BBI, της κοινή επιχείρηση. Θα κινητοποιηθεί λοιπόν, ελπίζω, ο προβλησμό από φέτο. Συνολικά δεν θα έχουμε αντίκτυπο επίπτωση στον συνολικό προπολογισμό. Και κάτι άλλο αφορά τις ε, επιχειρησιακές συνεισφορές σε ρευστό. Ούτε εδώ επηρεάζεται η κατάσταση. Δεν ε, αλλάζει το διοικητικό κόστος. Το 5% του κόστους του BBI πλέονται από την Κομισιόν και 50% το, από το BIC. Όπως είπε και κάποιος προλαλής σας, Προχωρούμε. Ευχαριστώ πολύ για τις φορέ σα. Ευχαριστώ τον κύριο Πόχα και όλους όσους ε, βοήθησαν. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Πόχα. Όλοι σα συγχαίρουν, ε, κύριε Πόχα. Τι λέτε. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, έχω το πλεονέκτημα να είμαι εισηγητής για τις οικονομικές δηλώσεις ε, για όλες τις κοινέ επιχειρήσεις. Είπαν πράγματι οι συνάδελφοι ότι έχουμε χαράξει το σωστό δρόμο. Ωστόσο, η, δια, δημόσια διαβούλευση μπορεί να μας δυσκολέψει ε, ακριβώς ε, γιατί μπορεί να επιβραδύνει τη διαδικασία από την οποία θέλουμε να ολοκληρώσουμε ε, εντός του 2018. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι επιχείρημα. Δεν είναι δυνατόν για αυτόν τον λόγο να μην γίνονται δημόσιες διαβουλεύσεις μήπως και εκφραστούν αρνητικές ε, απόψεις. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ο ιδιωτικός τομέας πριν από αρκετά χρόνια ήταν πρόθυμος να ε, αναλάβει αυτές τις δεσμεύσεις. Ίσως ε, τελικά ήταν μια παρεξήγηση αυτή που έγινε το 2014, διότι δεν κάνουμε έτσι τα πράγματα. Δεν αλλάζει τόσο γρήγορα ένας κανονισμός για κοινέ επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι έχουμε χαράξει το δρόμο προκειμένου να εγκριθεί ε, στη διάρκεια του φθινοπόρου και από εκεί και πέρα μπορούμε να ε, συνεχίσουμε τη διαδικασία το 2018. Ευχαριστώ πολύ. Εξ όσων θυμάμαι, βλέποντας ε, και την ε, ημερήσια διάταξη, πρέπει να σας πω ότι ήσασταν ο τελευταίος ομιλητής. Ε, προτού περάσουμε στα διάφορα, αν έχουμε διάφορα. Δεν βλέπω όμως κανένα να θέτει κάποιο θέμα. Επομένως θα τα ξαναπούμε στις 4 Σεπτεμβρίου. Να ευχηθώ σε όλους καλές διακοπές. Ο Πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς. Ευχαριστούμε και εμείς. Και τους ευχαριστεί για την πολύ καλή διερμηνία που προσέφεραν. Το είδαμε σήμερα και με, τους, με τις εστονούς υπουργούς. Και οι διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος, αξίζουν τις διακοπές τους. Και με αυτό ολοκληρώνουμε 40 λεπτά νωρίτερα. Κατά κάποιο τρόπο ξεπληρώνουμε το χρέος που έχουμε στους διερμηνείς από χθε που ε, δουλέψαμε 15 λεπτά παραπάνω και τους κρατήσαμε και εκείνους 15 λεπτά παραπάνω. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν στις 4 Σεπτεμβρίου. Γεια σας.